Uh, Καλημέρα. Και καλώς ήρθατε όλοι που ήρθατε εδώ για τη σημερινή μας ε, συζήτηση που θα κρατήσει λίγο πάνω από τρεις ώρες και θέλω να σας ενημερώσω ότι για να μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνάντησή μας αυτή. Να το ξέρετε. Λοιπόν, πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, την οποία την έχετε, γιατί έχει κυκλοφορήσει ήδη από την 3η 25 Απριλίου. Δεν ζήτησε κανείς καμία αλλαγή. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, σωστά. Οπότε εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Με ενημέρωσαν επίσης ότι πρέπει να κάνω μία ανακοίνωση, δεν είναι στην ε, ημερήσια διάταξη, και αυτό πριν περάσουμε στην ακρόαση. Θέλω να σας πω ότι από αυτή τη βδομάδα κάθε συνεισφορά στην νομοθετική διαδικασία από τα Εθνικά Κοινοβούλια είτε πρόκειται για τελογημένες γνώμες είτε οτιδήποτε στέλνεται στη διαδικασία αυτή νομοθέτησης θα είναι διαθέσιμες στο εσωτερικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο διαδίκτυο. Το λέω λοιπόν και για σας και για τους συναδέρφους σας από τα Εθνικά Κοινοβούλια να ξέρετε ότι ήδη από αυτή τη βδομάδα θα υπάρχουν όλες οι συνεισφορές σας εκεί. Και περνάμε στο δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι αυτό που ονομάζουμε για κοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη η συνάντησή μας αυτή στην εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης που αφορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας που ανέλαβε από την ΑΦΚΟ ο Παόλο Ράγκελ, ο συναδερφός μας, από το ΕΛΚ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι Πορτογάλος. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους μας εδώ που είναι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια από εννέα κοινοβουλευτικά σώματα από 8 χώρες μέλη είπαν ότι θα παρευρεθούν σήμερα εδώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε και το Διευθυντή Ενρίκο Φόρτη που είναι Διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σχέσεις μας με τα άλλα θεσμικά όργανα μεταξύ άλλων και τα κοινοβούλια. Σε λίγο θα του δώσω το λόγο. Προηγουμένως όμως, να συνεχίσω με το εξής. Ίσως γνωρίζετε ότι εδώ και χρόνια, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, έχουμε τέτοιες συναντήσεις της ΑΦΚΟ με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι πια παράδοση για μας. Συνήθως το Νοέμβριο έχουμε μια τέτοια συνάντηση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Πέρυσι, για παράδειγμα, ήταν το μέλλον της Ευρώπης το θέμα μας. Και σήμερα έχουμε μια έκτακτη τέτοια συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί εδώ και καιρό πιστεύουμε πως είναι αμοιβαίως εποφελές να έχουμε επαφές οι ευρωβουλευτές με τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε να συζητάμε μεταξύ μας. Στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα υπάρχει ρόλος για τα εθνικά κοινοβούλια αυτά καθεαυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα η ΑΦΚΟ ε, πιστεύει στον πολιτικό διάλογο και μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα της νομοθεσίας μας και αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί με συναντήσεις όπως είναι η σημερινή. Επίσης, για χρόνια έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτή την κοινοβουλευτική διάσταση και στις προηγούμενες θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε μάλιστα δύο εκθέσεις. Η μία ήταν του κύριου Καζίνη που ήταν πριν πρόεδρος της ΑΦΚΟ το 2014 και στη συνέχεια το 2009 ήταν του κύριου Μπρόκ. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια πάντως ήταν χρόνια εντατικού έργου και συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της ΚΟΖΑΚ για ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου ακριβώς, προκειμένου αυτός να γίνει πιο σταθερός, πιο μόνιμος και να αποτελέσει μια ισχυρή προστιθέμενη αξία. Μας βοηθούν σε αυτό και οι Βρετανοί συνάδελφοι θα έλεγα περισσότερο από ό,τι συνήθως. Συζητήσαμε την πρωτοβουλία για την πράσινη κάρτα, συζητήσαμε όλες τις πλευρές του διαρθρωτικού διαλόγου και μάλιστα κάποια εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν όχι μόνο στην ΚΟΖΑΚ αλλά και σε άλλες πλατφόρμες που έχουμε φτιάξει για την εξωτερική πολιτική, για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας, αλλά και για οικονομικά ζητήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε καλύψει όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και πιστεύουμε ότι από αυτή τη σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, εμείς, το Εθνικό Κοινοβούλιο, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην καλύτερη κατανόηση για το τι είναι η Ευρώπη ακριβώς. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε, αφού πρώτα μας ενημερώσει ο κύριος Ραγγελ για το περιεχόμενο της έκθεσής του και θα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε με τον κύριο Βάκλαφ Χάμπλα, πρώτα απ' όλα, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας της Τσεχίας. Στη συνέχεια, τον κύριο Βανίνο Τσίτη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από την Ιταλική Γερουσία. Δυστυχώς από τη Σουηδία δεν ήρθε ο συνάδελφος. Φαίνεται ότι έχασε το αεροπλάνο του. Τι να κάνουμε, συμβαίνει. Πού και πού. Και θα συζητήσουμε για την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης που αφορούν τα εθνικά κοινοβούλια. Και ο συνάδελφος από τη δικιά μας την πλευρά θα μας ενημερώσει και για το μέλλον των σχέσεων αυτών. Από πλευρά τώρα των εμπειρογνωμόνων υπάρχουν ε, κάποιοι που ήταν ευρωβουλευτές παλιότερα και που μας βοηθούν. Ε, ο κύριος Κάρλο Καζίνη για παράδειγμα που ήταν πρόεδρος της ΑΦΚΟ παλιότερα, θα μας μιλήσει για τη συνεργασία αυτή μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, τέος πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου της Πολωνίας, ο κ. Ντόν, που θα μας μιλήσει για την επικουρικότητα και έχουμε και τον Δ. Ίγκολφ Περνίτσε, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Χουμτόλ, που θα μας μιλήσει για τον πολιτικό διαφθρωμένο διάλογο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα, για τα πρακτικά. Πρέπει να περιοριστούμε όλοι σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. 10 λεπτά οι κύριοι ομιλητές. Οι άλλοι δεν υπάρχει όριο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να είσαστε σύντομοι. Σίγουρα πιο σύντομοι από 10 λεπτά. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Και μετά θα ακολουθήσουμε τη συνήθη παράδοσή μας, δηλαδή ένας ομιλητής από Εθνικό Κοινοβούλιο και ίσως δύο ευρωβουλευτές μετά, ανάλογα με την αναλογία που έχουμε. Συνήθως έτσι είναι. Αυτά είχα εγώ να σας πω εισαγωγικά. Ξαναθυμίζω, ξαναλέω ότι αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Ο κ. Φόλτ θα πάρει τώρα το λόγο για να μας μιλήσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των ε, και βουλευτέ από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρο Τίμερμαν ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί σα. Αύριο θα τον έχετε όμω, από ό,τι έχω καταλάβει, μαζί σα. Έχει οργανώσει μάλιστα και διάφορες συναντήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πολύ σύντομα, λοιπόν, εισαγωγικά, θέλω να σας πω ότι είμαστε στα μέσα του δρόμου, στα μέσα της θητείας της Ευρωπαϊκής αυτής Επιτροπής από τότε δηλαδή που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Γιούνκερ και όπου αφήνισε ότι οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια είναι πάρα πολύ σημαντική, μια από αυτοί βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Και μάλιστα η πρώτη πρόταση της έκθεσης του κύριου Ράγκερ λέει ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί χωρίς τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι αλήθεια. Όσον αφορά τώρα τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια έχει φανεί από την αρχή της θητείας μια που υπήρξαν πολλές επισκέψεις επιτρόπων που πήγαν ε, να επισκεφθούν τα εθνικά κοινοβούλια 500 μάλιστα ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε σε όλους τους επιτρόπους να φροντίσουν και να πάνε να επισκεφθούν τα εθνικά κοινοβούλια ε, πρόσφατα μάλιστα και επί τη ευκαιρία, το είπα αυτό, δηλαδή της κατάστασης πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο πρόσφατα το επανέλαβε όταν εγκρίθηκε η Λευκή Βίβλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια λοιπόν επίσης ετοιμάζουν πολλές συναντήσεις στο μέλλον για να ακούσουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις προτάσεις της για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι λοιπόν σημαντικό όχι μόνο να κρατήσουμε ψηλά τον πύχη για τη συνεργασία μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, βάσει των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει από τις ίδιες τις συνθήκες, αλλά και για έναν άλλον πολύ απλό λόγο. Ότι δηλαδή οτιδήποτε εγκρίνεται ως ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι κι πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, να εφαρμοστεί στις χώρες μέλη, άρα από τα εθνικά κοινοβούλια. Άρα λοιπόν αυτή η συνεργασία είναι στη φύση μας. Και όσο καλύτερη είναι η συνεργασία μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, τόσο καλύτερα θα εσωματωθεί και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην Εθνική. Βέβαια υπάρχουν και επίσημοι τρόποι, αλλά υπάρχουν και πιο ρεαλιστικοί τρόποι για να γίνεται αυτό. Ένας τρόπος είναι στο στάδιο προετοιμασίας του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την τελευταία φορά το 2016 και 2017 ο πρώτος αντιπρόεδρος απευθύνθηκε στα εθνικά κοινοβούλια ζητώντας τους απαντήσεις για αυτά τα οποία συνέβαιναν. Επίσης, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπονείται μια συγκεκριμένη στιγμή και τότε δίνονται πολλές ευκαιρίες στα Εθνικά Κοινοβούλια για επαφές ανάμεσα στην Επιτροπή και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ένας άλλος όμως τρόπος είναι πριν από την ενιαία πρωτοβουλία πριν διαμορφωθεί αυτή για τις αρχές της καλύτερης νομοθέτησης. Οποιαδήποτε νομοθεσία, οποιαδήποτε μάλλον νομοθεσίας προηγείται διαβούλευση με τον κόσμο. Και είναι και αυτή μια καλή στιγμή. Τώρα, για τα επίσημα τμήματα του πολιτικού διαλόγου. Θα υπάρξει μια έκθεση που θα εγκριθεί σύντομα τον Ιούνιο κατά πάσα πιθανότητα. Η έκθεση για τις ετήσιε δραστηριότητες με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εκεί θα δείτε ότι έχουμε όλο και περισσότερες νομοδοτήσεις που παίρνουμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πέρυσι ήταν 75%. Τεράστια αύξηση και είναι πολύ θετικό αυτό κατά τη γνώμη μας. Και πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ ό,τι γνωμοδοτήσεις παίρνουμε, είτε αιτιολογημένες γνώμες, είτε άλλες, φροντίζουμε και να απαντήσουμε πλήρως στο Εθνικό Κοινοβούλιο που μας έστειλε αυτή την γνώμη, όχι μόνο λόγω επικουρικότητας, αλλά και για οτιδήποτε άλλο και πιο τεχνικό μπορεί να περιλαμβάνει, να περιλαμβάνουν τα σχόλιά τους. Και δεύτερον, αυτό δεν το θεωρούμε εμεί σαν κάτι ερνητικό, ότι είναι για να μας τιμωρήσουν. Όχι, πιστεύουμε ότι έτσι βελτιώνεται πραγματικά η νομοθεσία μας. Τώρα, όσον αφορά την πράσινη κάρτα, δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί νομίζω ότι θα έχετε πολλές ευκαιρίες να το συζητήσετε. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι κάτι θετικό. Ότι είναι μια συνεισφορά των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ένα αρκετά νωρί στάδιο και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με δύο από αυτά. Μια που για μας η συνεισφορά αυτή είναι ιδιαίτερα θετική. Εδώ θα σταματήσω. Κατά τα άλλα, θέλω να σας ευχηθώ επικοδομητικό έργο. Και εμείς θα ακούσουμε όλες τις ιδέες που θα εκφράσετε και θα τις συζητήσουμε. Και ελπίζουμε και εμείς να έχουμε πάντα καλό και καρποφόρο διάλογο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Πάολο Χανζέολ που είναι ο λόγος ε, της συγκέντρωσης όλων σας εδώ μαζί μας. Πάολο, έχεις το λόγο όχι πάνω από 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Καταρχά, θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω όλο, όλα τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που συμμετέχουν ε, σήμερα και τον κύριο Βάκλακ Χάμπλ και τον κύριο Βανίνο Κίτη όλος ιδιαιτέρως που θα αναπτύξουν τα θέματα αυτά αλλά και τον πρώην Πρόεδρο και πολύ καλό φίλο Κάρλο Καζίνη καθώς και τον κύριο Λούτβιχ Ντόρν και τον καθηγητή Ίγκολφ Πέρνιτσε που για μένα είναι ε, πέρα από πανεπιστημιακός και ευρωπαϊκή αναφορά για το θέμα αυτό. Τώρα θέλω να πω ότι έχω μια κάποια εμπειρία σε αυτό το ζήτημα διότι στην τελευταία θητεία ήμουν αντιπρόεδρος του ΕΛΚΑ αρμόδιος για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Συμμετείχα λοιπόν επανειλημμένα στις ε, συνεδριάσεις της ΚΟΖΕΑΚ και άλλες συνεδριάσεις ε, που συμμετείχαν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και ασχολούνταν με το θέμα αυτό και θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς επίσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ακόμη περισσότερο όμως ανάμεσα στις δύο διαστάσεις των κοινοβουλίων, τα εθνικά με το ευρωπαϊκό. Ορισμένε φορές τείνουμε να πιστεύουμε πως υπάρχει ένα είδος θεσμικής ζήλιας ε, ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το ε, εθνικό επίπεδο, ειδικά ε, όσον αφορά τα κοινοβούλια. Όμως η αλήθεια είναι ότι η δημοκρατική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται απολύτως από τη συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά και το Ευρωκοινοβούλιο καθώς και από τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι εάν συνεργαστούμε θα έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικό έλεγχο στο έργο της εκπροσώπησης των λαών μας και γι' αυτό είναι σημαντικό να δημιουργηθεί αυτό, αυτή, το πνεύμα αγαστής συνεργασίας. Εδώ λοιπόν σε αυτό το προπαρασκευαστικό κείμενο έχουμε θέσει στην ουσία κάποιες ερωτήσεις και περιμένουμε να λάβουμε, όπως ήδη είχαμε σε κάποιες επαφές που έχουμε ήδη ξεκινήσει, τις δικές σας συμβολές για αυτά τα ζητήματα. Φυσικά θα έλεγα ότι το πρώτο θέμα, το οποίο είναι το πιο δημοφιλές θα έλεγα, είναι το θέμα της ε, επικουρικότητας. Να κατανοήσουμε δηλαδή ακριβώς πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον έλεγχο της ε, επικουρικότητας πώς θα μπορέσουμε να συντονίσουμε και να οριστικοποιήσουμε τις εθνικές ε, από τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και επίση να δούμε κατά πόσο αυτός ο έλεγχος της ε, επικουρικότητας θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και το συνομοσπονδιακό ε, ζήτημα. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό ας πούμε. Να θίξουμε και το, το θέμα δηλαδή της, της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο και πώς θα γίνει αυτό. Έπειτα, θα πρέπει να δούμε αυτές τις 8 ή 12 εβδομάδες αν τις παρατείνουμε στο μέλλον όπου τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους και να έχουν και πρόσβαση στις μεταφρασμένες εκδοχές, γιατί κάποιες φορές η επικοινωνία δεν διευκολύνεται διότι δημοσιεύεται ας πούμε αυτό που αποφασίζουν, αλλά δημοσιεύεται μόνο στην εθνική γλώσσα. Οπότε τα υπόλοιπα κοινοβούλια έχουν δυσκολίες. Τεχνικές δηλαδή ε, πτυχές, ε, οργανωτικές πτυχές που όμως είναι πολύ σημαντικές ώστε να δημιουργούνται οι ευκαιρίες για διάλογο ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια για να μπορούν και εκείνα να παρεμβαίνουν ε, σε εθνικό επίπεδο. Επίσης άλλο θέμα είναι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και εδώ πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Ενρίκο Φόρτη και τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς που έδωσαν ε, πολύ μεγάλη προσοχή στα θέματα που μας απασχολούν. Η πρωτοβουλία Μπαρόζο αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο και είναι σαφές ότι ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαντς είναι απόλυτα προσιλωμένος ε, ε, στην εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων για τα ευρωπαϊκά, στα με τα ευρωπαϊκά θέματα. Στη συνέχεια. Αυτό που νομίζω ότι είναι κάπως νέο γιατί η ιδέα της έκθεσης δεν είναι μόνο να γίνει κάποια αξιολόγηση, ένα είδος ε, στατιστικής για τα βήματα που έχουν ήδη γίνει, αλλά θέλουμε και να σκεφτούμε και να προβλέψουμε πώς θα βελτιωθεί αυτή η σχέση. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσουν δύο-τρία ε, ζητήματα. Το πρώτο που είναι αρκετά σημαντικό είναι τι είδους συνεδριάσεις θα πρέπει να οργανώσουμε και με ποια σώματα Ποια είναι η εξολόγηση που κάνουμε για την εργασία της ΚΟΖΑ και, και μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα πιο αποτελεσματικό. Επίσης μια άλλη πολύ παλιά πρόταση που την έχω όμως υποβάλει μόνο σε επίπεδο ΕΛΚ είναι να οργανώσουμε ένα είδος ευρωπαϊκής ομάδας όπου δηλαδή ταυτόχρονα το Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα αφοσιώνονται στη μελέτη των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ας πούμε παρουσία των ευρωβουλευτών στη Εθνικά Κοινοβούλια και όχι μόνο ευρωβουλευτών από την ίδια χώρα αλλά και από άλλες χώρες εκπρόσωποι τη Κομισιόν, εν πάση περιπτώσει μια εβδομάδα όπου ταυτόχρονα σε όλα τα κοινοβούλια θα συζητώνται ευρωπαϊκά θέματα και όπου θα μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε έναν απολογισμό του έτους για τα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτή είναι μια πρόταση. Μετά έχουμε την πράσινη κάρτα και την κόκκινη κάρτα. Ε, ιδιαίτερα η πράσινη κάρτα θα πρέπει να διερευνηθεί, δηλαδή η δυνατότητα ε, που θα δοθεί έτσι στα εθνικά κοινοβούλια να, να μπορούν να αναλάβουν κάποιο είδους πρωτοβουλίας Δηλαδή κάτι που έχει ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορούν να υποβάλουν αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ασκήσει ή τουλάχιστον να υποχρεωθεί να εξηγήσει γιατί δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της, την πράσινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα δε, θα πρέπει να είναι μια άλλη ε, δυνατότητα ή μια ευκαιρία. Και τέλος κάτι ακόμα που πιστεύω ότι είναι σημαντικό, να αναπτύξουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποιος, ε, κάποια άρθρα των καταστατικών των Εθνικών Κοινοβουλίων, των κανονισμών συγγνώμη, των Εθνικών Κοινοβουλίων, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά στην εξέταση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Και να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Κάποιες φορές ορισμένοι εθνικοί βουλευτές ανησυχούν γιατί λένε ότι χάνουν αρμοδιότητες σε δημοσιονομικά θέματα λόγω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τι συμβαίνει λοιπόν. Σε πορά από τα Εθνικά Κοινοβουλία το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σχεδόν το αγνοούν. Ε, εξακολουθούν να ακολουθούν τις παλιές διαδικασίες για τον προϋπολογισμό. Εάν όμως γίνει η συζήτηση για του Γενικού προϋπολογισμού πριν από την υποβολή του πρώτου εγγράφου από την Εθνική Κυβέρνηση στις Βρυξέλλες, το Εθνικό Κοινοβούλιο αν δηλαδή προβλέψουμε, αν κάνουμε ένα είδος εθνικού εξαμήνου, εθνικού τριμήνου πριν από το ευρωπαϊκό εξάμεινο, πολλές πολύ μεγάλο μέρος της δυνατότητας επιρροής και της δυνατότητας λήψης αποφάσεων των εθνικών κοινοβουλίων θα ανακτηθεί πλήρως. Άρα λοιπόν, με κάποιες πρωτοβουλίες που μπορεί να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μικρές αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Βεβαίως, καθένα από αυτά είναι, ε, κυρίαρχα να το αποφασίσουν ή όχι. Πάντως, θα μπορούσαν να παίξουν πιο δραστηριό ρόλο συμμετέχοντας σε αυτού του είδους της πρωτοβουλίας. Και έτσι αυτή η αίσθηση, η εντύπωση απώλειας κυριαρχίας θα μπορούσε έτσι να ξεπεραστεί γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο στην πράξη να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τον εθνικό χρόνο με τον ευρωπαϊκό χρόνο, να συγχρονίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τις εργασίες, ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν μια πολύ πιο ε, στεναρή παρουσία στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Όλες αυτές οι προτάσεις και ερωτήσεις είναι στο προπαρασκευαστικό έγγραφο και γι' αυτό και ε, περιμένουμε να ακούσουμε τις δικές σας συμβολές και να ενισχύσουμε τον διάλογο για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και γραπτό τους επόμενους μήνες πριν να ε, κρίνουμε το σχέδιο έκθεσης. Σα ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα εδώ ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Πάολο. Θα περάσουμε τώρα στον κύριο Βάτσλαβ Χάμπλ, που είναι από την Γερουσία της Τσεχίας, πρώτος ομιλητής από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Dear Chair, dear... Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. εγώ ε, θα χρησιμοποιήσω την τεχνολογία που μας προσφέρετε. Θα με βλέπετε στην οθόνη. Δυστυχώς θα έχω την πλάτη μου γυρισμένη σε όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τον κύριο Ραγγέλ, Ραντζέλ για, την, για τα σχόλιά του και επίσης και για την πρόσκληση που μας απίπτυνε να πούμε και εμείς τη γνώμη μας με βάση το τι κάνουμε στη γερουσία της Τσεχίας και το τι συζητήσαμε τους τελευταίους μήνες ε, στην Επιτροπή της Γερουσίας για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα από αυτά που θα ακούσετε είναι δικά μου σχόλια. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στην Τσεχία η Γερουσία έχει διαφορετικό ρόλο από την Κάτω Βουλή. Την Βουλή των Αντιπροσώπων, των Βουλευτών. Συγκεκριμένα, η γερουσία δεν έχει πολλές αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού. Αυτά ρυθμίζονται περισσότερο από το Κοινοβούλιο, από την Κάτω Βουλή. Ως εκ τούτου, τα θέματα αυτά θα ήταν καλύτερα να τα ακούσετε από κάποιον βουλευτή της κάτω βουλής. Εγώ θα κάνω απλώς ακροθυγός κάποια σχόλια. Θα ήθελα επίσης να τοποθετηθώ σε αυτά που ελέγχθησαν με βάση αυτά που διαδραματίζονται στη δική μας Γερουσία. Δηλαδή οι συζητήσεις σε εμά για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικότητα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι κάθε άλλο. Εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα την πολύ καλή δουλειά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δεν, δεν θέλουμε να αναλάβουμε εμείς κάποιες από τις αρμοδιότητές του. Το βασικό μας κίνητρο είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προσπαθούμε δηλαδή ε, να βελτιώσουμε την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον το πώς την εκλαμβάνει η κοινή γνώμη. Γιατί στην Τσεχία αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας. Δηλαδή οι Τσέχοι πιστεύουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει λιγότερη δημοκρατική νομιμοποίηση από αυτή που πραγματικά ε, υπάρχει. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ βασικό κίνητρο, δηλαδή να βελτιώσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα ήθελα να σχολιάσω σύντομα και τα διάφορα θέματα της ερωτήσεις που ετέθησαν ε, στο προκατρακτικό έγγραφο. Ε, Τίθε το θέμα του ελέγχου της επικορικότητας. Συζητήσαμε για το ρόλο της συμμόρφωσης με την αρχή της επικορικότητας, ότι αυτό αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, πολιτικούς φορείς. Δεν πρόκειται για έλεγχο νομιμότητας. Η αντίδραση των ε, εθνικών κοινοβουλίων πρέπει να γίνει αποδεκτή Δεν πρόκειται για αυστηρά οριζόμενη επικουρικότητα, αλλά έτσι την αποδίδουμε με ευρύτερη έννοια και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, και ο έλεγχος ε, της επικουρικότητας δεν πρέπει να ερμηνεύεται με την στενή έννοια, γιατί αναμφίβολα δεν σημαίνει κανένα απολύτως κίνδυνο για την νομοθετική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθεί σε εμά να μην υπάρχει το δικαίωμα της αρνήσης κυρίας. Ε, δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε νομοθεσία. Αν θέλετε μπορούμε να καθυστερήσουμε. Ναι, αυτό ναι. Αλλά σε τελική ανάλυση Ίσως μπορούμε να επιφέρουμε και κάποιες βελτιώσεις για το πώς πρέπει να γίνονται τα διάφορα νομοθετικά βήματα στα κράτη-μέλη. Εγώ πιστεύω ότι ο έλεγχος επικουρικότητας πρέπει να περιλαμβάνει και έναν έλεγχο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν έλεγχο της νομικής βάσης. Διότι Εάν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν νομική βάση για να αντιδράσουν, είναι λογική συνέχεια ότι δεν μπορεί και να εκπληρώνεται η αρχή της επικορικότητας, η οποία είναι συνειφασμένη με την ε, ε, νομική βάση. Τα εθνικά κοινοβούλια, ακόμα και αν θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αναλογικότητα. Ε, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σωστό ε, και νόμιμο, ηθικό και νόμιμο να προβληθεί αυτό το θέμα στα επιχειρήματα και στις ε, γνωμοδοτήσεις που έχουν σχέση με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Δεν πρέπει δηλαδή να δίνουμε σημασία μόνο στην αναλογικότητα. Και κάτι άλλο, και δεν νομίζω βέβαια ότι ε, σας λέω κάτι το καινούριο, ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τον έλεγχο της επικουρικότητας είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια πολλές φορές είναι απογοητευμένα γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία ε, θετική επίπτωση από αυτά που διαδραματίζονται. ένα εθνικό κοινοβούλιο σίγουρα σε επίπεδο αρχή δεν μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Παρ' όλα αυτά όμως ε, πρέπει να υπάρχει ε, να είναι πιο σαφείς οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Αυτό θα βελτιώσει την αποδοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτά που λέω δεν ε, σημαίνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία. Αλλά θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένε επιπτώσεις, έστω και μικρές, να παρουσιάζονται, να εξηγούνται, να γίνονται κατανοητές. Και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί βέβαια η αντίδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τουλάχιστον σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά παρόλα αυτά ε, θα είναι πολύ καλύτερα αν το επίπεδο της ε, επιχειρηματολογίας εξετάζοντας συγκεκριμένες ε, αντιδράσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων αν βελτιωθεί η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν στο προκαταρκτικό έγγραφο υπάρχει και μία τεχνική ερώτηση σχετικά με την επέκταση ε, του χρόνου για τον έλεγχο της επικουρικότητας, να φτάσει δηλαδή ε, περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα, το καινούριο χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει και νομίζω ότι θα βελτιώσει και πάρα πολύ ε, τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ε, σας είπα ήδη, νομίζω ότι αυτά που ισχύουν ε, για τον έλεγχο επικορικότητας ισχύουν και για τον πολιτικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίως όσον αφορά στις αντιδράσεις της Επιτροπής. Μερικές φορές οι αντιδράσεις δεν είναι πολύ συγκεκριμένες και η Επιτροπή πολλές φορές επαναλαμβάνει τα προηγούμενα επιχειρήματα. Οι επιπτώσεις ε, από αυτά που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απόλυτα σαφείς. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρονται με μεγαλύτερη σαφήνεια. Όσον αφορά την πράσινη κάρτα, νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, ε, κυρίως και πάλι για να βελτιωθεί η ύπαρξη ή η έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης. Μέχρι τώρα πιστεύω ότι όλη η διαδικασία είναι ικανοποιητική. Βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια προόδος με αυτές τις ε, κοινέ πρωτοβουλίες με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να παρουσιάζονται νέες πολιτικές, ε, να παρουσιάζονται αποτελέσματα. Εάν λοιπόν υπάρχει καλή, ε, υπάρχει θέληση και αυτά μπορούν να λειτουργήσουν στο μέλλον. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει πάρα πολλές απόψεις για την πράσινη κάρτα και ίσως τα πράγματα να συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον το στοιχείο της ε, καλής θέλησης ε, για την ύπαρξη αυτού του μηχανισμού, αυτό το στοιχείο είναι πιο σημαντικό από το ίδιο το στοιχείο και το περιεχόμενό του. Όσον αφορά την κόκκινη κάρτα. Εδώ πρέπει να σας πω, ε, κυρίως μετά το Brexit, πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς όπως υπήρχε και πριν από την αξιότητα της Μεγάλης Βρετανίας Το γεγονός λοιπόν ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί μια τέτοια κόκκινη κάρτα, νομίζω ότι αυτό θα βελτιώσει το πώς ε, οι πολίτες ενός κράτους μέλους ε, αντιμετωπίζουν ε, νομοθετικές πράξεις που θα μπορούσαν να αναχαιριστούν από ε, πολίτες άλλων κρατών μελών. Αν όχι να, να σταλούν, ε, να οδηγήσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξανασκεφτεί ε, πολλά θέματα. Θέλω να σας πω ότι θα μου άρεσε να εξεταστούν όλα αυτά. Η κόκκινη κάρτα ως σχεδιάστηκε πριν από το δημοψήφισμα για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας είχε ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ο αριθμό των εθνικών ε, κοινοβουλίων που θα έπρεπε να συμμετέχουν ήταν, ε, λέγε, 55 άτομα τουλάχιστον περισσότερο δηλαδή από ότι η μειονότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου τα εθνικά κοινοβούλια καταρχήν έχουν την δύναμη να ε, δρομολογήσουν αυτή την κόκκινη κάρτα, ακόμα και αν συμμετέχουν λιγότερα κοινοβούλια. Ε, πάντως πιστεύω ότι το να υπάρχει ένας τέτοιος στάνταρτ μηχανισμός, αυτό νομίζω ότι έχει κάποια αξία. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν αναθεωρήσουμε τις συνθήκες, κάτι που νομίζω αυτή τη στιγμή κανείς δεν το επιθυμεί. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν αυτή τη δυνατότητα και δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αναθεωρήσουμε, να ξανανοίξουμε δηλαδή το θέμα των συνθήκων. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των μειονοτήτων στα εθνικά κοινοβούλια, Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και μειονότητες να καταθέτουν την άποψή τους. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα. Αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσον ε, θα χρησιμεύσει και θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί ακόμα και για σημαντικές γνωμοδοτήσεις δεν βλέπουμε να υπάρχει ε, μεγάλη δραστηριότητα γιατί δεν έχουν και επιπτώσεις, δεν έχουν συνέχεια αυτές οι γνωμοδοτήσεις. Καλή ιδέα των μειονοτήτων. Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάποιο βαθμό όλα αυτά ήδη γίνονται. Παραδείγματος χάνει στη δική μου τη χώρα. Διότι οι δύο βουλές που έχουμε εμείς έχουν και πολιτικά τελείως διαφορετική σύνθεση γιατί εκλέγονται με διαφορετικούς μηχανισμούς, με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν ε, το κοινοβούλιο ε, κατ' ουσίαν είναι, έχει περισσότερο πολιτική χρειά, διότι ε, τα κόμματα που έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ορίζουν και την κυβέρνηση. Στη Γερουσία τα πράγματα είναι διαφορετικά και εκεί ίσως και απόψη Γερουσίας να αποκλίνουν λιγάκι από αυτές του Κοινοβουλίου. Αυτό έχει σημασία και ίσως κάπου να παρουσιάζεται και στα έγγραφα. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι παΐων επί του θέματος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενδεχομένως ε, να ε, εμπλέκεται με σημαντικές ε, οικονομικές πολιτικές μιας χώρας, Υπάρχει πράγματι κάποια αρμοδιότητα των κρατών μελών και ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά και εδώ το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αλλά καθαρά πρακτικά ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν αρκετό χρόνο για να μπορούν να συζητάνε ε, το σχέδιο συστάσεων πριν αυτές οι συστάσεις εγκριτούν από το Συμβούλιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η νυν Επιτροπή προσπαθεί να το πράξει και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Φαντάζομαι δεν έχω πια άλλο χρόνο. Είχα κι άλλα να πω, αλλά θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάμπλου. Ο κύριος Βανινοτσίτη από το Ιταλικό, από την Ιταλική Γερουσία. Παρακαλώ. Κύριε Κίτη, έχετε το λόγο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Χούμπνερ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Ρανζέλ, για, καθώς και τα μέλη της ε, <clears throat> Επιτροπής ε, τη Συνταγματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή σα την πρόσκληση, ώστε να κάνουμε μια την παραβολή των προποθέσεών μα ε, για αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάνω από 7 χρόνια έχει μπει σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα και είναι σωστό να συνεχίσουμε και να βαθύνουμε ε, της, ε, το προβληματισμό μας για το τι ακριβώς σημαίνει η πρόβλεψη του άρθρου 12 της συνθήκης με βάση το οποίο τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, σε αυτή την κατάσταση ακριβώς όπου βρισκόμαστε με το δημοψήφισμα που αποφάσισε τον αποχωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολιτικές δυνάμεις που ως στόχο έχουν την έξοδο από την από το ευρώ και από την ίδια την Ένωση και με θέματα διεθνών σχέσεων που δεν είναι τώρα ε, στιγμή να σας θυμίσω ε, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της ε, Ιταλικής Γερουσίας, η συνεργασία, συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της, των ιδεωδών της Ευρώπης, αλλά και για την οικοδόμηση μιας προόδου προς αυτή την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναφερθεί πρόσφατα στην ε, Σύνοδο στη Ρώμη για την 60η επέτειο ε, των συνθήκων. Ελευθερία, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλεγγύη είναι οι πυλώνες που γέννησαν, που διέπουν και που θα συνεχίσουν να ε, επιτρέπουν την πρόοδο στην Ένωση. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα λειτουργήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό. Εγώ καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων στον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γιατί ξεκίνησε με τον πολιτικό διάλογο. Είναι ένα, δηλαδή μια επί της εξέταση των ευρωπαϊκών θεμάτων ε, σε μια σχέση πρώτα της Κομισιόν με τα Εθνικά Κοινοβουλία που οδήγησε και στην ευάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτή η προσπάθεια ήδη ευνόησε μια μεγαλύτερη διάδοση. Αν σκεφτώ ότι γινόταν πριν από 5-10 χρόνια, μεγάλη διάδοση των περιεχομένων των δραστηριοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου στα, ανάμεσα στους, τους πολίτες μας. Πολλές ε, επιτροπές της Γερουσίας ασχολούνται με ευρωπαϊκά θέματα στις δραστηριότητε τους και κυρίως η Πολιτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, θα ήθελε να ε, μπορεί να εκδίδει μια προληπτική γνωμοδότηση για τη συνοχή με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Ε, τα εθνικά κοινοβούλια μπόρεσαν έτσι να παρακολουθούν πολύ πιο ενήμερα τις δραστηριότητες των ίδιων τους των κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί σε πολλά κοινοβούλια όπως και στο δικό μας πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρος της κυβέρνησης έρχεται και ε, κάνει μια ενημερωτική παρουσίαση για τις θέσεις που θα προτάξει. Δίνουμε λοιπόν εμείς κάποιες κατευθύνσεις και 15 μέρες, εντός μάλλον 15 ημερών από τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέ, οφείλει να έρθει και να ενημερώσει. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίζουμε με μεγάλη διαφάνεια τι ακριβώς συμβαίνει στις ε, δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έπειτα αυτό βοήθησε και σε, μια καλύτερη, σε ένα καλύτερο συντονισμό των διαφόρων διατάξεων στις διάφορες χώρες. Τώρα, ε, το Ιταλικό, η Ιταλική Γερουσία εξ αρχής πίστεψε σε αυτήν την συνεργασία και θα εξετάσει επί της ουσίας τις προτάσεις. Ε, όχι μόνο δηλαδή τις δικές, αυτές τις οποίες περιλαμβάνονται στο έγγραφο του εισηγητή Ρανζέλ. Θα εξετάσουμε εις βάθος τις προτάσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δική μας συμβολή, γιατί είναι σήμερα σημαντικό να εντατικοποιηθεί ο διάλογος με το Ευρωκοινοβούλιο, ακριβώς έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή ε, πορεία. Μια άλλη φορά όταν είχα έρθει στην Βρυξέλλας είχα συνομιλήσει με τον υπεύθυνο του Κοινοβουλίου και είχαμε στηρίξει αυτήν τη στάση, δηλαδή ε, θέλαμε να στηρίξουμε και κάτι νέο που εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, δηλαδή νομοδοτήσεις, ψηφίσματα και τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια αποτελούν τμήμα του φακέλου συνεδρίασης της Επιτροπής. Αυτός δηλαδή είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος για να ενισχυθεί η συνεργασία στην ουσία της νομοθετικής διαδικασίας και πιστεύω πως ε, από αυτή την άποψη όπως μας προτείνει και ο εισηγητής, πιστεύω πως είναι χρήσιμο να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερες διμερείς ε, ανταλλαγές ανάμεσα στους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για αυτά τα θέματα όπου θέλουμε να, ε, να, να εντατικοποιηθεί η συνεργασία και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, ε, ιδιωτικό και ζωή, υγεία, περιβάλλον, μετανάστευση κτλ. Η Ιταλική Γερουσία και μαζί και με άλλα κοινοβούλια συμμετείχαμε στα πρώτα σχέδια ε, και τις προτάσεις για το πράσινη ε, κάρτα, για την ε, περιβαλλοντική ευθύνη, την εταιρική ευθύνη, είδα και τον συνάδελφο που το πρότεινε και έχουμε σε αυτό προσιλωθεί με μεγάλη πεποίθηση. Και αυτό το οποίο αξιοποίησε ακόμη περισσότερο αυτό το θετικό μέσο δημοκρατικής συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων ήταν ότι το ορίσαμε ως ε, ενισχυμένο πολιτικό διάλογο. Αυτή η φάση, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να παραμείνει άτυπη, χωρίς να της δώσουμε δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μορφή, αλλά αυτό το θέμα της πράσινης κάρτας καλό θα είναι να αναπτυχθεί, γιατί είναι ένας θετικός τρόπος ε, ώστε να μην μπλοκάρονται οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, να συμβάλλουμε στο να κάνουμε κόμμα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να υπερασπιστούμε κοινά μας ε, project και ε, συμφέροντα εγώ αντίθετα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της Τσεχίας είμαι αντίθετος με την κόκκινη κάρτα ωστόσο γιατί τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με τη συνθήκη συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία της Ένωσης και άρα λοιπόν κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια προσέγγιση που σημαίνει επικοδομητικό ρόλο ενώ η κόκκινη κάρτα έχει αρνητικό χαρακτήρα δηλαδή ε, στην ουσία είναι τιμωρητικό η ακυρωτική η λειτουργία της ε, κόκκινης κάρτας. Για μένα θα πρέπει να ε, τονίσουμε τον ε, πολιτικό διάλογο, την αντιπαράθεση, τη γόνιμη ε, θα μπορούσε να υπάρχουν κοινοβούλια που να είναι αντίθετα με τις ευρωπαϊκές προτάσεις και από αυτών των αξιολογήσεων το Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, τα ευρωπαϊκά, καλό θα είναι ένα ναι εμβαθύνων. Αλλά πιστεύω πως το δικό μας κοινό συμφέρον των ευρωπαϊστών είναι να συμμετέχουμε και όχι να μπλοκάρουμε τις διαδικασίες λήψης απόφαση. Ε, ε, το ίδιο ακριβώς το, το λέω και για τον μηχανισμό ελέγχου της, αλληλη, της επικουρικότητας. Αυτό βοήθησε πολλά εθνικά κοινοβούλια να εξετάσουν ευρωπαϊκά ζητήματα, όμως παραμένει ένα μέσο με περιορισμένες δυνατότητες Μεταξύ άλλων έχει ερμηνευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρει περιπτώσει, το κίτρινο, η κίτρινη κάρτα ω ένα μέτρο για να στηριχθούν περισσότερο οι εθνικέ θέσει των εθνικών κυβερνήσεων και όχι πραγματικά ω καταγγελία τη παραβίαση τη αρχής της επικουρικότητας. Και έπειτα, εάν δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ή εν πάση περιπτώσει αν κενωθεί από την ουσία του, αυτό ε, έγινε λόγω του μηχανισμού που προβλέπεται στο πρωτόκολλο νούμερο 2 αλλά και μάλλον κάτι που ξεχάσαμε, κάτι που, στο οποίο θα πρέπει να προσυλλοθούμε περισσότερο να αποφασίσουμε να δώσουμε βάρος σε αυτό το, ανακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, να υπάρχει ένα είδος ε, γραμματείας για τα πιο σημαντικά θέματα όπου θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε την κίτρινη κάρτα. Για μένα όμως ε, πιο σημαντικό είναι και επαναλαμβάνω είναι ο πολιτικός διάλογος. Επιπλέον θεωρώ ότι οι συνθήκες σήμερα δεν διευρύνουν, δεν προβλέπουν μάλλον την επέκταση των αρμοδιοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων στον έλεγχο της νομιμότητας ούτε στον ε, ε, έλεγχο της αναλογικότητας. Αν δεν υπάρξει σχετική απόφαση του δικαστηρίου ε, θα είναι να μείνουμε στην προστιθέμενη μόνο αξία ε, που έχουμε με βάση τις παραμέτρους ε, λειτουργίες που εν γέννη αναγνωρίζονται. Τελε, προτελευταία μου παρατήρηση είναι αυτή που αφορά το πείραμα των επιτροπών, ε, στις οποίες ήδη αναπτύσσονται εδώ χρόνια, αναπτύσσεται μάλλον εδώ και κάποια χρόνια συνεργασία ανάμεσα στα Εθνικά και το Ευρωκοινοβούλιο. Και αναφέρομαι πέρα από την Κόζα, την οποία δεν αναφέρατε κι εσείς, τη ε, σύσκεψη ΠΕΣ και ΠΕΣΔΕ, τη διάσκεψη για τα προβλήματα του προπολογισμού, την Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από τους Προέδρους των ε, Κοινοβουλίου. Εδώ νομίζω είναι ένα πρόβλημα και πρέπει και αυτό να το σκεφτούμε. Πόσο δηλαδή αυτές οι επιτροπές που ήδη είναι ένα μέσο με μια συνέχεια συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, το Εθνικά Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό, πώς θα μπορέσουν να είναι αναφορά για την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων αντιπροσωπεύουν, που αντιπροσωπεύονται από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τώρα, στο μια λογική συνεργασία, αυτό που δεν είναι ο πυρήνα ε, ενό ε, τρίτου σώματος, ε, κοινοβουλευτικού σώματο Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο δεν θα έχει νόημα. όμω η εταιρική αυτή σχέση θα μπορούσε να είναι σημαντική, ώστε η εκμεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου να μπορεί να έρχεται σε επαφή με του βουλευτέ των κρατών μελών για να αντιμετωπίζουν τα σημαντικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάμεινο με το εξάμεινο. Ας πούμε τώρα η Μάλτα, η Προεδρία της Μάλτας, αυτό το οποίο προτάσει είναι εμβάθυνση στα θέματα της μετανάστευσης στην Μεσόγειο και εκεί συμμετέχουν εθνικοί βουλευτές από πολλά κράτη-μέλη και το αποκορύφωμα θα είναι αυτή την εβδομάδα στη Σικελία ε, για να συζητήσουν τις δυσκολίες, το περίπλοκο χαρακτήρα διαχείρισης ενός εποχικού φαινομένου που δεν μπορεί παρά να ενδιαφέρει κάθε Ευρωπαίο πολίτη και κυρίως έτσι ώστε να επαληθευτεί η συνέπεια και η συνέχεια ανάμεσα στις αξίες ε, της αλληλεγγύης, της προτεραιότητας, της αξιοπρέπειας του ανθρώπου με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα επί των οποίων έχει γεννηθεί και αναπτυχθεί η Ένωση και να δούμε όλα τα ε, πήγοντα περιστατικά που διαδέχονται το ένα το άλλο. Τέλος, ε, ναι, η, μια τέτοια συμφωνία δεν θα λύσει. Δεν θα δώσουμε τώρα απαντήσει σε όλα τα προβλήματα, ότι θα λύσουμε όλα, αλλά συμφωνώ. Με τα όσα είπε ο, ο, ο εισηγητή ε, Ρανζέλ, ότι δηλαδή θα πρέπει να διοργανώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα ευρωπαϊκών θεμάτων σε όλα τα κοινοβούλια, ώστε μαζί με τους εθνικούς βουλευτές να έρχονται και, και ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της Κομισιόν. Γιατί κάτι το οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε είναι ότι ανάμεσα στα όσα συζητώνται στις επιτροπές για τα ευρωπαϊκά θέματα, στις ειδικές επιτροπές, οι σχέσεις με τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δυνατότητα συμμετοχής του Ευρωκοινοβουλίου είναι αυτά που συζητώνται περισσότερο. Νομίζω λοιπόν πως αυτή η πρόταση θα μπορούσε να προχωρήσει συγκεκριμένα. Τελευταίο θέμα αφορά, κατά τη γνώμη μου, τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στα θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εδώ έχουμε πολύ κρίσιμα ζητήματα γιατί διάφορα άρθρα της συνθήκης δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν. Αν σκεφτεί κανείς τους κανόνες που ισχύουν για τους μηχανισμούς αξιολόγησης των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών για τα θέματα δικαιοσύνης εσωτερικών υποθέσεων, τους μηχανισμούς ε, σύνδεσης και αξιολόγησης της δραστηριότητα του Eurojust, ο πολιτικός έλεγχος του Europol, άρθρα 70, 85 και 88. Πιστεύω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια οφείλουν Θέλω να θέσουν ως στόχο την ανάκτηση αυτής της, την κάλυψη μάλλον αυτής της μεγάλης καθυστέρησης και να βρουν διαρθρωμένες μορφές συνεργασίας ώστε να είναι εγγυημένα τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών γιατί εν τέλει όταν μιλάμε για συνεργασία στην ε, νομοθετική διαδικασία και σχέση συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, το κεντρικό ζήτημα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Τα δικαιώματα των πολιτών που πάνω απ' όλα ε, έχουν, ε, μάλλον αντιπροσωπεύονται από το Κοινοβούλιο και ζητούν ακριβώς από τα κοινοβούλια μια κοινή συνεργασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της προοπτικής στην Ευρώπη. Ε, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, Γερουσιαστή κύριο Κίτη. Πάμε τώρα στους εμπειρογνώμονες και θα ήθελα να έχετε καλοσύνη να μιλάτε 10 λεπτά για να μπορούν και άλλοι συνάδελφοι να ε, λάβουν το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Καζίνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η δική μου παρέμβαση βασίζεται στην ε, έκθεση την οποία έχω συντάξει για αυτή την επιτροπή. Τη συνέταξα βέβαια στην προηγούμενη θητεία, αλλά αναφέρομαι ε, και σε άλλες εκθέσεις του 97, 97 και μέχρι σήμερα και εκθέσεις άλλων συναδέλφων, των συναδέλφων Απολιτάνο και Μπρόκ. Έχουν παρουσιαστεί λοιπόν όλε αυτές οι εκθέσεις στην ΚΟΖΑΚ ε, και στην προηγούμενη θητεία είχαμε κάνει συζητήσει με όλα τα εθνικά κοινοβούλια για να μπορέσουμε πολύ ελεύθερα και χωρίς δυσκολίες χρόνου να ακούσουμε τις απόψεις των κοινοβουλίων επ' αυτών των ε, θεμάτων. Έτσι λοιπόν ε, Υπάρχει αναμφίβολη κρίση. Η κρίση για να ξεπεραστεί πρέπει να υπάρχει και αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και να σα εξηγήσω γιατί πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικά Κοινοβούλιο. Αυτό είναι δεσμευτικό, είναι παγιωμένο ε, και στη συνθήκη τη Λισαβόνα ε, και στι καταμέρου συνθήκε. Όμω ε, πρέπει να σα πω εγώ με απασχόλησε πάρα πολύ αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 12 τη συνθήκη τη Λισαβόνα, όπου αναφέρεται ότι τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά στην εύρυθμη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ενεργά, τι ακριβώ σημαίνει, ε, από ό,τι φαίνεται, τα εθνικά κοινοβούλια δεν ε, είναι ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να δίνουν και ένα κίνητρο για την ε, περαιτέρω ολοκλήρωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστική σημασία. Είναι κάτι το οποίο κατ' ουσίαν όμως ε, θέτει να αμφιβόλω όλη αυτή την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει πλήρης ολοκλήρωση. Στη συνθήκη της Λισαβόνας, στο άρθρο 11, μιλάμε για μια φάση που είναι μια φάση ενδιάμεση με ένα συγκεκριμένο στόχο και μια συγκεκριμένη πορεία. Επ' αυτού όμως οι ιδρυτικές συνθήκες δεν λένε τίποτα. Λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ε, πιο ενωμένη, πιο αυστηρή. Άρα δηλαδή είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η διαδρομή ε, θα πρέπει να είναι δημοκρατική. Εάν όμως τελικά το σχέδιο είναι να υπάρχει μια πολιτική ένωση ομοσπονδιακής μορφής, νομίζω ότι αυτό είναι διαφορετικό από την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένα δίκτυο που θα συνδέει διάφορα κράτη-μέλη και θεσμούς. Η δημοκρατική αρχή είναι σαφές, απαιτεί αυτό που σήμερα ονομάζεται δεύτερη βουλή, δηλαδή το Συμβούλιο να έχει μια δημοκρατική, μεγαλύτερη δημοκρατική έκφραση. Θα μπορούσε να υπάρχει μια ερετή δεύτερη βουλή που θα προέρχονται οι εκλεγμένοι ερετοί από τα κράτη-μέλη. Αν από την άλλη θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα, έχει απλά ένα δίκτυο διασύνδεσης και τίποτα άλλο, τότε τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει ε, να μπορούν να αποστασιοποιούνται από την ευρωπαϊκή αυτή εκπροσώπηση. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο, επί το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή η δημοκρατική αρχή απαιτεί και προϋποθέτει αυτό που εμείς μιλάμε εδώ για την δεύτερη βουλή, το Συμβούλιο να είναι εκείνο που να εκφράζει τη δημοκρατική τέληση των λαών. Γιατί ε, το να ελέγχουν τα κοινοβούλια τους υπουργούς, αυτό είναι απολύτως απαραίτητο πρέπει λοιπόν στα κράτη-μέλη, στην Ιταλία συγκεκριμένα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νόμος. Θα πρέπει λοιπόν στα κράτη-μέλη να προβλέπετε ότι η συζήτηση προηγείται και ακολουθεί προφανώς συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ε, ακολουθεί και και ακολουθεί μετά από το, ε, τις συναντήσεις ε, του Συμβουλίου των Υπουργών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 2009 που ε, για την συνθήκη της Λισαβόνας είπε ότι η Ευρωπαϊκή, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να πρέπει να νομιμοποιείται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έτσι ώστε οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση των αρμοδιοτήτων να απαιτεί την επιβεβαίωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχω ήδη παραθέσει από τον Ιταλικό νόμο που προσπαθεί να κωδικοποιήσει λιγάκι αυτό τον ε, διάλογο ανάμεσα στο ε, στα Κοινοβούλια και το Συμβούλιο, όπου το Συμβούλιο εκφράζει περισσότερο τη λαϊκή βούληση. Για μένα το σηκότερο όλων είναι ότι το συνταγματικό αρχιτεκτόνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη τα κοινοβούλια ε, και για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή συνείδηση. Αυτό είναι πολύ απαραίτητο αν θέλουμε να πλησιάσουμε τους πολίτες και για να ενισχύσουμε τα αισθήματά τους ότι ανήκουν στην ίδια την Ευρώπη για να ξεπεράσουμε τους ε, εθνικισμούς και να μπορέσουμε να βαδίσουμε προς την ολοκλήρωση. Εδώ λοιπόν τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν ε, δυνατότητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό λοιπόν εγώ κατά το παρελθόν μίλαγα για αντεστραμμένη επικουρικότητα Υπάρχουν πράγματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να τα κάνουν μόνο τα Εθνικά Κοινοβούλια και αυτό αφορά κυρίως στην ευρωπαϊκή, στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Συνείδησης. Σύντομα λοιπόν ε, θα ήθελα να πω κάτι ίσως ε, και για την κόκκινη κάρτα που για να τεθεί αυτό ε, σε λειτουργία πρέπει να υπάρχει νομίζω 95, υπογραφή 95 ευρωβουλευτών. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Πιστεύω ακριβώ το αντίθετο γιατί δημιουργεί σύγχυση και τελικά θα πρέπει να υπάρχουν χαρακτηριστικά μιας τρίτης ε, βουλής ε, που εγώ το αποκλείω. Άρθρο 12 σχετικά με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Νομίζω αυτά τα έχω ήδη πει. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας ε, κατάλογος συγκεκριμένων εργαλείων συνεργασίας ε, να είναι εργαλεία προκαταρκτικά ε, πριν υπάρχει κάποια δέσμευση και όλα αυτά να συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο. Ε, γιατί και αυτή η συνάντησή μας μπαίνει σε μία συνάντηση των θεσμών Και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τις συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η ΚΟΖΑΚ υπάρχει από το 89 και στην Κόζακ, όπως ξέρετε, μάλλον η Κόζακ, όπως ξέρετε, συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Οι πρόεδροι της Κόζακ ε, συμμετέχουν βέβαια και σε πολλές άλλες συνεδριάσεις για να υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση όλων των απαραίτητων εργαλείων. Η ε, διακοινοβητική συνέλευση που βασίζεται στο άρθρο 13 του Συμφώνου Σταθερότητας αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων όπως προβλέπεται και στο συνθήκη της Λισαβόνα, άρθρο 88 αναφέρθηκε προηγουμένως στην Πρατισλάβα οι πρόεδροι των Κοινοβουλίων πρόσφατα αποφάσισαν να συστήσουν μία ε, συνδιάσκεψη σε επίπεδο Europol. Νομίζω ότι πρέπει να διοικηθούμε. Αρκούν όλα αυτά ή πρέπει να υπάρξουν και άλλα. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να ε, δημιουργηθούν ε, άλλα εργαλεία. Υπάρχουν φιλόσοφοι αρχαίοι οι οποίοι λένε ότι δεν χρειάζεται να δημιουργούνται άλλοι θεσμοί αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Θα ήθελα σύντομα να μιλήσω για την Κόζα, γιατί αυτή με ενδιαφέρει πάρα πολύ κατά το παρελθόν. Υπάρχει εδώ το θέμα της ταυτότητας της Κόζακ. Δεν αρκεί να λέμε ότι ε, δεν μπορούμε να καταργήσουμε την Κόζακ γιατί προβλέπεται από τις συνθήκες. Πρέπει να δώσουμε όμως ένα χρήσιμο σκοπό. Το έχω πει και στην προηγούμενη θητεία, ο στόχος θα μπορούσε να είναι έτσι πολύ ευρύτερος, δηλαδή η Κόζακ να ελέγχει ε, το τι έχει γίνει σε όλες αυτές τις εκφάνσεις της, ε, των προσπαθειών ε, για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσω για τον έλεγχο της ελεκτρονικότητας, γιατί θα μιλήσει όποιος ακολουθήσει μετά από εμένα. Πιστεύω όμως ότι ε, αυτό που ελέγχθη για την πράσινη κάρτα. Εγώ ανέκαθεν πίστευα ότι ο έλεγχος της επικουρικότητας, ε, κατά την άποψή μου, ε, δεν έχει σχέση άμεση με το να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες τις, που έχουν σχέση με την αναλογικότητα. Άρα δηλαδή εδώ σαφώς αυτή η πράσινη κάρτα μπορεί άμεσα τη σχέση με την αναλογικότητα. Πάντως η επικουρικότητα δεν πρέπει να είναι τροχοπέδι. Τουναντίον θα πρέπει να είναι ε, εργαλείο συνεργασίας, δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια και τύχη ακόμα και αν ε, τα, οι κάρτες ε, από τότε που συστήθηκε αυτό το δημόσιο υπήρξαν μόνο τρεις, παρόλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές ε, παρατηρήσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Περίπου 400 ε, αιτιολογημένες ε, γνωμοδοτήσεις, οι επιτροπές τα έχουν μελετήσει όλα αυτά και ας μην ξεχνάμε ότι το άρθρο 12 της συνθήκης ζητάει από τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετέχουν όπως είπαμε ενεργά. Άρα δηλαδή ίσως θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οποτεδήποτε φτάνει κανείς σε ικανοποιητικό επίπεδο συμφωνίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, θα μπορούν να λαμβάνεται υπόψη η δική τους η άποψη σε περίπτωση αδράνειας της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτό μπορεί κανείς ε, να πλησιάσει στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν τότε τα αντίστοιχα κοινοβούλια να υποβάλουν την, προσ... την πρόταση. Η Κόζακ θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη έδρα για την εκτίμηση των πράσινων και κίτρινων καρτών, καθώς και εκείνων των προτάσεων που δεν έχουν ακόμα οριμάσει αρκετά, πριν ε, δηλαδή να πάρουν τη μορφή πράσινης κάρτας στο πλαίσιο της Κόζακ. Ωστόσο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό πρόβλημα. Δεν φαίνεται να μπορούμε να σκεφτούμε δεσμευτική επίπτωση της πράσινης ε, κάρτας, ώστε δηλαδή ό,τι προτείνει να γίνεται κατευθείαν ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία. Αντίθετα, θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίση, κάτι ακόμα πιο σοβαρό προκύπτει. Το θέμα της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα φαίνεται πως τελείω ε, την έχουμε εμπιστευτεί στην Κομισιόν. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι πολύ αμφισβητήσιμος κανόνας γιατί σε κάθε κυβέρνηση οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα της πρωτοβουλίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να, αναρωτηθούμε για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών που θα πρέπει να προετοιμαστεί με βάση μια απλή αναφορά και τελικά να μην αν δεν οδηγεί σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, τότε καλύτερα να το καταργήσουμε και τελείω. Και αυτό είναι μια πρόταση, κάτι που λέω σε σχέση με γενικά τι αναφορέ. Χρειάζεται ωστόσο μια εμβάθυνση δημοκρατική στο θέμα της πρωτοβουλίας. Να μπορεί η πρόταση να απορριφθεί, αλλά να μπορεί και να βρεθεί συμβαστική, που θα ορίζει ότι η Κομισιόν θα λειτουργεί ως φίλτρο, ως χώρος αναδιατύπωσης και αναθεώρησης. Αν όμως θέλουμε να δώσουμε πρωτοβουλία στο Εθνικά Κοινοβούλιο, δεν θα έπρεπε να δώσουμε στη ε, Κομισιόν τη δυνατότητα διαγραφής ή κατάργησης μιας πρότασης. Περιορίστηκα λοιπόν σε αυτά τα ολίγα για να μπορέσουν και οι άλλοι δύο εμπειρογνώμονες να αναπτύξουν περισσότερο τα άλλα τους θέματα, αλλά θα κάνω και μια παρατήρηση που αφορά την σχέση ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Εθνικό Κοινοβούλιο και τα ε, πολιτικά κόμματα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή θα εντοτικοποιηθεί η σχέση εάν υπάρξουν αυθεντικά πολιτικά κόμματα ευρωπαϊκού επίπεδου όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 214 της, ε, του Οκτωβρίου σε σχέση με το, στατο, το καταστατικό της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Αυτά τα ευρωπαϊκά κόμματα που είναι παρόντα και στα εθνικά κοινοβούλια θα έπρεπε να ευνοήσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα εθνικά κοινοβούλια, να κινητοποιήσουν σε ευρωκοινοβούλιο με πιστικό τρόπο το σεβασμό των απόψεων των Εθνικών Κοινοβουλίων να ορίσουν ενωτικές στρατηγικές γραμμές καθώς και να φτιάξουν και ένα σύστημα διακυβουλευτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία των ίδιων των πολιτικών κομμάτων μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κατά κάποιο τρόπο να διέπονται με από κάποιου κανόνες ή διακοινοβουλευτικέ συναντήσεις των κομμάτων που ήδη γίνονται. Οι τελευταίε ευρωεκλογέ. ε, είχε προταθεί από τα ίδια τα κόμματα, είχαν προταθεί μάλλον οι συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, επίσης θα μπορούσε να υπάρξει μια διεθνής, ε, διεθνή ψυχοθελτία, αλλά εδώ υπάρχουν δύο πτυχές. Εγώ δεν εκφράζω τη δική μου γνώμη, λέω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν αυτά τα ζητήματα. Αυτή την... Ε, ο διεθνή χαρακτήρα ενό ε, τόσων βουλευτών είναι πολύ περίπλοκη. Δεν φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Όμως θα απελευθερωθούν θέσει με το Brexit, έδρες μάλλον θα πρέπει ίσως αυτές να δοθούν σε μια διεθνή, ένα διεθνές ψηφοδέλτιο. Θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτό το λέω γιατί όπως είπαμε πρέπει να εντατικοποιηθούν και να τονιστούν οι σχέσεις μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Τώρα. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λούτβικ Ντόρνο που ήταν πρόεδρος στην Πολωνική Βουλή. Θα μας μιλήσει για την επικουρικότητα και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με το εξή. Μου είπαν ότι πρέπει να σας μιλήσω για την επικουρικότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα ήθελα ευθύ εξ αρχής να καταλήξω στο εξή συμπέρασμα. Ότι για την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή από τη μία και τα Εθνικά Κοινοβούλια από την άλλη, η αρχή της επικουρικότητας και οι μελέτες σχετικά με την επικουρικότητα βάζουν κάποιους περιορισμούς. Και για να το πω διαφορετικά. Τι μπορούμε να πετύχουμε υπέρ της Ευρώπης. Μέχρι τώρα σίγουρα έχουμε πετύχει πολλά χάρη σε αυτή τη διαδικασία η κίτρινη κάρτα για την επικουρικότητα. Έχουμε πετύχει ήδη πολλά. Αυτό λοιπόν που πρέπει τώρα να θέσουμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω για αυτή την αρχή της επικουρικότητας που μπαίνει βέβαια στις σχέσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με τα εθνικά κοινοβούλια. Να δούμε λοιπόν πώς αυτές οι σχέσεις μέσω της επικουρικότητας μπορούν να γίνουν πιο στενές. Σε αυτό θα καταλήξω. Αλλά θέλω τώρα να αναφερθώ σε τρεις περιπτώσεις τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η κίτρινη κάρτα για να δούμε ποια είναι η γλώσσα και ποια είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν τα Εθνικά Κοινοβούλια και ποια είναι η απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μελετώντας λοιπόν την κατάσταση διαπιστώνουμε ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ίδια την αρχή της επικουρικότητας, έχει να κάνει περισσότερο με πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή για τα εθνικά κοινοβούλια, τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό είναι κάτι το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα μέσα από το μηχανισμό της κίτρινης κάρτας. Και πρέπει αυτό να διατυπώνεται σε μία γλώσσα που να είναι κατανοητή για τη χρήση της επικουρικότητας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι ολοφάνερο και προβλέπεται από την ίδια τη συνθήκη. Σήμερα δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις, υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο τι λέμε και τι υπάρχει στο περιεχόμενο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, ότι υπάρχει δηλαδή μια απόκληση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Δεύτερον, όσον αφορά τον περιορισμό των ελέγχων, όσον αφορά την ε, διαδικασία της επικουρικότητας και πώς τη χρησιμοποιούν τα εθνικά κοινοβούλια. Εδώ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν παραδέχεται, γιατί ποτέ δεν μπορεί να το παραδεχτεί, αλλιώς θα είναι σαν να αρνείται τις ίδιες τις, τις εξουσίες. Αρνείται λοιπόν ότι έχει πάει πιο μακριά από την αρχή της επικουρικότητας ενώ πρέπει να είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Και ω θεματοφύλακα των συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πώ είναι δυνατόν να παραδεχτεί ότι έχει ξεπεράσει τι εξουσίε τη. Με άλλα λόγια, αν έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Εθνικά Κοινοβούλια δίκιο έχετε, τότε είναι σαν να αυτοκυρώνεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν μια κατάσταση, ένα φοβερό παράδοξο Κανείς που έχει το μυαλό του στη θέση του δεν θα αντιδρούσε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, στα πλαίσια πάντα της αρχής της επικουρικότητας και πώς ασχολούμαστε με αυτή την αρχή. Ο έλεγχος της αρχής της επικουρικότητας μας οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα μηδέν. Δηλαδή, ή που γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας ή δεν γίνεται σεβαστή και κάποιος ξεπερνάει τις αρμοδιότητες του. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια ε, θα κερδίζει και αυτοί που χάνουν είναι τα εθνικά κοινοβούλια. Άρα εδώ δημιουργείται μονίμως μια φοβερή απογοήτευση. Αυτές είναι οι αρχές σχετικά με τις οποίες πιστεύω ότι με τις παρατηρήσεις του συγητή πρέπει να μας προβληματίσουν και να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτές. Δηλαδή η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Για την αναλογικότητα δεν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Η αρχή της αναλογικότητας είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει την εφαρμογή μιας πολιτικής με δημοκρατικό τρόπο. Υπάρχει δηλαδή αυτό το αντιστάθμισμα, το αντίβαρο. Διότι αν όλοι υποχωρούν υπερβολικά, τελικά κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Οπότε αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα μείνουμε λιγότερο δυσαρεστημένοι. Είναι η σύγκριση ανάμεσα στην αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κανονικά θα έπρεπε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο μιλητή για να ε, πει τα δικά του ζητήματα, αλλά δύο θέματα θέλω να θίξω ακόμα στα δέκα λεπτά που μου δώσατε. Και είναι τα εξή. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι το εξή. Διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, Αν δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην αρχή της αναλογικότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να είναι το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο το περισσότερο δυνατό. Αυτό δηλαδή που θα σταμάταγε την απομόνωση των εθνικών κοινοβουλίων όπου αυτή υπάρχει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φαίνεται πολύ ομή, αλλά στην πραγματικότητα έχει μία ιεραρχική δομή σαν αυτοκρατορία. Στις αυτοκρατορίες υπάρχει το σύστημα της ρόδας που γυρίζει, χωρίς όμως να ξέρουμε ποιο είναι το κέντρο. Στα Εθνικά Κοινοβούλια διαπιστώνουμε ότι η ακτίνα της ρόδας, η οποία δηλαδή συνδέει το κέντρο με την περιφέρεια έχει ενισχυθεί. Και αυτό είναι καλό. Υπάρχουν λοιπόν νέα συμφέροντα τα οποία αναδύονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μια μισορροπία για να μην υπάρχουν αδιέξοδα, γιατί στην ε, αναλογικότητα μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν υπάρχει ποτέ αδιέξοδο. Πώς θα χειριστούμε λοιπόν την επιρροή του κέντρου, ώστε να έχουμε ακόμα και συγκρούσεις, οι οποίες όμως να είναι επικοδομητικές, να καταλήγουν σε κάτι θετικό και να μην είναι καταστροφικού τύπου. Αν καταφέρει κανείς να δαμάσει μια σύγκρουση και την χρησιμοποιεί επικοδομητικά, μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας, να θεωρήσουμε ότι η σύγκρουση αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για να λύσουμε τις διαφορές μας. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Οι ακτίνες της ρόδας είναι αυτές οι οποίες κάνουν τη ρόδα να γυρνάει. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Το κέντρο από μόνο του δεν φτάνει. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ και σας, κύριε Ντόν, για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις σας. Θα έχουμε συζήτηση και σίγουρα πολλοί θα αναφερθούν σε αυτήν. Τώρα, η τρίτη παρέμβαση είναι του καθηγητή Ίγκολφ Περνίτσε. που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Humboldt, που θα αναφερθεί στον δομημένο ε, διάλογο, τον πολιτικό δομημένο διάλογο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω γερμανικά, λέει ο μιλητής. Βεβαίως. Είναι καλό, λέει ο μιλητής, ακόμα και για τους διερμηνείς. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Ράγκελ για τις ερωτήσεις που μας έστειλε και οι οποίες πραγματικά μπαίνουν στο κέντρο του προβληματισμού μας. Το πρώτο που θα κάνω είναι να εκφράσω μια προειδοποίηση. Η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές δεν λειτουργεί αρκετά καλά επειδή δεν ξέρουμε ποιος είναι αρμόδιος γιατί. Όταν λοιπόν μιλάμε για έναν δομημένο πολιτικό διάλογο, αυτό ακριβώς είναι που μπορεί να βοηθήσει, γιατί έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου να μπερδεύεται ακόμα περισσότερο το πράγμα για το ποιος είναι αρμόδιος γιατί. Και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε Ποιο είναι υπεύθυνο γιατί και να εντοπίσουμε ποιο δεν κάνει καλά τη δουλειά του και ποιο την κάνει καλά. Πώς μπορούμε λοιπόν εκείνοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ε, να αναγκαστούν να λογοδοτήσουν. Το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο. Εάν τώρα ε, απευθυνθούμε σε όλα τα κοινοβούλια και τους πούμε ότι κοιτάξτε εσείς θα είσαστε υπεύθυνοι για όλα ε, και θα αποφασίζετε ε, τότε δεν ξέρω τι ακριβώς θα, προθείς, τι θα προκύψει. Αυτό που έχει σημασία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία για να υπάρχει και δημοκρατική νομιμοποίηση. Επιτρέψτε μου μία πρώτη γενική παρατήρηση. Για μένα ισχύει το εξής. Διαπιστώνουμε ότι στα κράτη-μέλη ε, κυρίως ο ρόλος των ε, εθνικών κοινοβουλίων δεν ακολουθεί τις πραγματικές εξελίξεις. Δηλαδή, ε, τα εθνικά κοινοβούλια, το γιατί υπάρχουν, αυτό δεν ακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Πολλά ε, πολιτικά θέματα που αφορούν στους πολίτες, αν ισχύει ότι αυτά κρίνονται στις Βρυξέλλες και αν ισχύει επίσης αυτό που λέει το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το άρθρο 10 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούνται στα, ε, στο Συμβούλιο ε, είναι, οφείλουν να λογοδοτούν απέναντι στα κοινοβούλια. Αν ισχύει αυτό, τότε και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σε προεκλογικές εκστρατείες, σε εθνικά, σε κράτη-μέλη, γιατί σε αυτές τις ε, προεκλογικές εξαρτίες τα ευρωπαϊκά θέματα κατ' ουσίαν δεν παίζουν κανένα απολύτω ρόλο. Κανένα απολύτως ρόλο. Η Καλσουρουή το νότιο συνταγματικό δικαστήριο, λέει ότι οι Βρυξέλλες έχουν αποφασίσει για πάρα πολλά θέματα, όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν παίζει κανένα απολύτω ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες οι κυβερνήσεις ε, που λαμβάνουν τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες, κυρίως ε, το Συμβούλιο που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές. Μα ποιος ελέγχει το Συμβούλιο, μόνο τα Εθνικά Κοινοβούλια, δεν υπάρχει κανένας άλλος και ως εκ τούτου υφίσταται το εξής πρόβλημα, ότι Πρώτα απ' όλα πρέπει αυτό να το συνδυτοποιήσουν τα εθνικά κοινοβούλια και αφού το συνειδητοποιήσουν θα λαμβάνουν πιο σοβαρά υπόψη τους ε, τις ε, υποχρεώσεις τους και έτσι θα υπάρξει και πολύ καλύτερη συνεργασία γιατί η εκτελεστική εξουσία, η Κομισιόν και το Συμβούλιο χρειάζονται ε, ισχυρό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, εγώ θεωρώ ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργάζονται στενά. Περνώ τώρα σε μία τρίτη προκατρακτική παρατήρηση. Πρόκειται για την αρχή της ε, επικουρικότητας. Και στην αρχή της επικουρικότητας υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις. Η αρχή της επικουρικότητας εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο των εθνικών κοινοβούλιων κατά της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής, κατά της ε, ευρωπαϊκής υπερεξουσίας στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι παρανόηση. Η επικουρικότητα είναι ένα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προϋπόθεση της νομοποίησης ευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, το ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται εκείνα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ή να γίνουν αποτελεσματικά στα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου, ε, προκύπτει επιπρόσθετη αρμοδιότητα και δραστηριοποίηση προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Και η αρχή της ε, επικουρικότητας είναι η αρχή εκείνη η οποία ρυθμίζει το τι πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά πόσον ε, θα πρέπει να λειτουργεί κανείς προδραστικά και όχι με τη μορφή της υπεράσπισης της Ευρώπης. Πόσο λοιπόν μιλάμε για το σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης, προφανώς και μιλάμε για την προστασία των εθνικών αρμοδιοτήτων έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν η πράσινη κάρτα είναι μια πολύ καλή σκέψη. Θα πρέπει πράγματι να σκεφτούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια μεταξύ άλλων έχουν το καθήκον να σκέπτονται ποιους στόχους επιθυμούν να επιτύχουν. Και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν σε Εθνικό Κοινοβούλιο μόνο, άρα χρειάζονται την Ευρώπη ως εκ τούτου. Τα Εθνικά Κοινοβούλια στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το πολύτιμο εργαλείο που είναι η Ευρώπη για να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να ε, προστατεύσουν καλύτερα τους πολίτες τους. Με αυτήν λοιπόν την ερμηνεία της αρχής της επικουρικότητας νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε αυτές τις θαυμάσιες δέκα ερωτήσεις του κυρίου Ράγκελ και το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση. Εγώ θα αναφερθώ και στις 10 ερωτήσεις. Πρώτο ερώτημα. Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση επ' αυτού του θέματος. Παράδειγμα, η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κυρίου Τόιφελ στην ε, διακυβερνητική, ο οποίος ε, προσπάθησε να πάρει πίσω τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν τον ρώτησαν, μα ποιες, είπε τελικά δεν βρέθηκε καμία να είναι υπερβολική. Και ο κύριος Κάμερον και αυτός το προσπάθησε με την περίφημη αναθεώρηση της ισορροπίας των αρμοδιοτήτων. Πίστευε ο κύριος Κάμερον ότι είχε βρει ένα θαυμάσιο όπλο έναντι της Ευρώπης. Τελικά αυτό αποδείχθηκε ολοκληρωτική καταστροφή για τον κύριο Κάμερον, αλλά νίκη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σε αυτή την έκθεση που προετοιμάστηκε δεν αναφέρθηκε ούτε μία αρμοδιότητα που να κρίθει ότι περισσεύει και ότι είναι υπερβολική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου αυτή η συζήτηση καταπίπτει. Πάμε στο δεύτερο, στο σύστημα της ε, έγκαιρης ε, προειδοποίησης. Πράγματι δεν είναι αποτελεσματικό. Μπορούμε αν θέλετε να συζητήσουμε για τις προθεσμίες. Εγώ δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον ε, μεταγενέστερη προθεσμία ή διορία ε, θα βελτιώσει αυτό το σύστημα της ε, έγκυρης προειδοποίησης. Εντάξει, ενδέχεται να αναλυφθούν κάποιες περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλά εγώ πιστεύω και μόνο η ύπαρξη αυτής, εγω πιστευω και μονο η υπαρξη αυτου του συστήματος και η αρχή της επικουρικότητας με έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καταθέτει νομικές πράξεις αντίθετες προς την επικουρικότητα. Βέβαια, θα μπορούσαμε το σύστημα αυτό να το καταστήσουμε αποτελεσματικότερο με την έννοια ότι θα μπορούσαμε να προβάλλουμε και να συμπεριλάβουμε στο σύστημα την ιδέα των μειονοτήτων. Πρώτα απ' όλα, μπορεί κανείς να ερωτήσει γιατί μία ομάδα κρατών να μπορούν να ε, προκαλέσουν αυτό το σύστημα της έγκυρης προειδοποίησης. Αν όμως πρόκειται για ομάδα κρατών μελών, τότε πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν και διαφορετικές ισορροπίες. Ε, δεν είναι ίδιες παντού οι ισορροπίες τις περισσότερες φορές ε, τα κοινοβούλια στην πλειοψηφία του συμμορίζουν την κυβέρνηση και δεν θα αμφισβητήσουν την κυβέρνηση. Αν πούμε ότι χρειαζόμαστε έναν, ε, μια υπερκομματική συμμαχία αν θεωρήσουμε ότι χρειαζόμαστε κάποια κοινοβούλια και κάποιες μειονότητες από άλλα κοινοβούλια να συνέλθουν όλοι αυτοί, ας πούμε να πούνε οι σοσιαλιστές αυτό δεν γίνεται ή οι συντηρητικοί να πούνε ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Κομισιόν γιατί παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, τότε ενδεχομένως οι συνεργασίες που ε, προκύπτουν μέσα από τις συμμαχίες, αν γινόντουσαν όλα αυτά, θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε περισσότερη πολιτικοποίηση της Ευρώπης. Και αυτό το χρειάζεται η Ευρώπη, την πολιτικοποίησή της. Να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτής της πολιτικοποίησης, ποιες είναι οι θέσεις που υπάρχουν για την ανεργία, για την πολιτική λιτότητα. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και ίσως με ένα ε, τέτοιο σύστημα έγκυρης προειδοποίησης να τα καταφέρουμε όλα αυτά καλύτερα. Περνάω στην πράσινη κάρτα και αυτή θα μπορούσε να είναι οργανωμένη με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ένα κοινοβούλιο ή μια συμμαχία μια συγκεκριμένη πολιτική ε, κατεύθυνση από διάφορα κοινοβούλια να αναλάβει μια πρωτοβουλία έναντι τη Κομισιόν. Και αυτή είναι μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν χρειάζεται μια διάταξη στη συνθήκη για να γκρίνει κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν τέτοιες πρωτοβουλίες από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μα είναι σαφές ότι αν πούνε κάποιες ομάδες από Εθνικά Κοινοβούλια στην Κομισιόν σας παρακαλούμε Κομισιόν κάντε μια πρόταση για αυτό το θέμα προφανώς και η Κομισιόν θα πρέπει να καταθέσει πρόταση και έτσι να προχωρήσει η Ευρώπη. Αν θέλετε, η Κομισιόν πρέπει να έχει πιο ανοιχτά τα αυτιά της, να στραφεί περισσότερο προς τα κοινοβούλια και τους πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πολιτικοπούσε αν θέλετε, περισσότερο την κατάσταση και θα την έφερνε πιο κοντά στον πολίτη. Περνάω τώρα στον πολιτικά διαρθρωμένο διάλογο. Αυτό τώρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε του κυρίου Μπαρόζου. Να το αναγνωρίσουμε ότι αυτό ξεκίνησε από το 2006. Έκτοτε συνέβησαν πάρα πολλά. Αντιλάγησαν πάρα πολλά έγγραφα, έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Έχω ένα βιβλίο εδώ, όπου ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο κύριος Γιάν Κούπα, σε αυτό το βιβλίο του για τα Εθνικά Κοινοβούλια μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και την κρίση της Ευρώπης, αν κατάλαβα καλά τον συγγραφέα και αν καταλαβαίνω καλά αυτά που ακούω από εδώ και από εκεί, αυτές οι επιτροπές και η συνεργασία μεταξύ τους. Πολύ ωραία όλα αυτά. Γνωρίζονται οι άνθρωποι, τα συζητάνε, τα λένε πάρα πολύ ωραία. Όμως φαίνεται ότι ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικό να δουλεύουν στην εκλογική τους ε, περιφέρεια και όχι να συμμετέχουν ε, σε αυτούς τους ε, διαλόγους. Και όλα αυτά μοιάζουν να σχετίζονται με το ότι αυτοί, αυτές οι διάφορες επιτροπές της κοινοβουλευτικής συνεργασίας, αυτές δεν έχουν καμία αρμοδιότητα λήψη απόφασης, τίποτα. Λένε κάτι, αποφασίζουν κάτι, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτές τις αποφάσεις. Τουλάχιστον, ε, εγώ δεν διαβάζω τίποτα για όλα αυτά στις εφημερίδες. Δεν ενημερώνεται η κοινή γνώμη. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον είναι λογικό και απαραίτητο να εκχωρήσουμε έστω κάποιες αρμοδιότητες λήψη αποφάσεων σε αυτά τα φόρουμ, σε, αυτά, σε αυτούς τους οργανισμούς. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση της συνθήκης για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω τρεις βασικής, βασικοί τομείς ε, όπου μπορούν να υπάρξουν όλα αυτά είναι το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Εκεί ε, γίνονται και λέγονται πάρα πολλά, αλλά η αρμόδια επιτροπή δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις. Το δεύτερο, ε, στην, στην πολιτική εξωτερικών και άμυνας και εκεί γίνονται συζητήσεις. Δεν λέω τώρα ότι οι συζητήσεις ε, είναι περιτές, αλλά λέω ότι αν υπήρχε αρμοδιότητα λήψη αποφάσεων αυτής ε, της ε, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Αν υπήρχε αυτό, τότε οι υπουργοί και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, θα έτειναν περισσότερο ευήκο για να ξέρουν τι γίνεται. Και θα ενισχύεται στην περίπτωση αυτή η κοινοβουλευτική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνώ στη Europol, Joint Scrutiny Committee για τη Europol αυτοί ίσως να έχουν κάποιες ε, σημαντικές αρμοδιότητες λήψη αποφάσεων, δεν το γνωρίζω. Αν το έχουν, αυτό όμω θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τις άλλες επιτροπές. Πάω στο επόμενο θέμα, στην πράσινη κάρτα ναι, κόκκινη κάρτα όχι και να σας πω γιατί η κόκκινη κάρτα για μένα δεν είναι σωστή. Υπάρχει μια θεσμική ισορροπία υπάρχει μια διάταξη του πώς τρέχουν οι αρμοδιότητες και πού βρίσκονται οι ευθύνες. Η κόκκινη κάρτα λοιπόν αυτό το θέμα της ε, ευθύνης και της λογοδοσίας θα το ανακάτευε, θα το ανέτρεπε Ίσως κάποια κοινοβούλια να το βρίσκουν αυτό πολύ ελκυστικό, το να μπορούν να βγάλουν κόκκινη κάρτα. Όμω ο πολιτικό έλεγχο για αυτά που διαδραματίζονται στις Βρυξέλλε μετά από πρόταση τη Κομισιόν του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, η πολιτική ευθύνη βρίσκεται σε αυτού του θεσμού και αυτοί οι θεσμοί λογοδοτούν η Κομισιόν στο Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσει στα εθνικά του κοινοβούλια. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία και μια κόκκινη κάρτα απλά θα δημιουργούσε ένα ρήγμα. Άκουσα προηγουμένως τη λέξη αναταραχή και εγώ έτσι το βλέπω. Θα το θα δημιουργεί το πρόβλημα στο σύστημα και ε, δυστυχώς υπάρχει κίνδυνο στο το σύστημα να ετίθετο ένα αμφιβόλο. Πάω στο εργαλείο IPAX. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο είναι μια βάση ενημέρωσης και επικοινωνίας για την διακοινοβουλευτική συνεργασία. Απαραίτητο λοιπόν εργαλείο για να ενισχυθεί η συνεργασία αυτή και διαρωτώ με κατά πόσον στο πλαίσιο του IPAX μπορεί να υπάρχει και κάτι που θα άγγιζε την όλη συζήτηση για τα ε, τις πλατφόρμες συζήτησης online. Δηλαδή, όταν γίνεται ε, διακοινωτική συνεργασία για συγκεκριμένα θέματα, αυτή η συνεργασία αποκτά νόημα μόνο εφόσον ad hoc επιλαμβάνεται κάποιων θεμάτων και δεν ε, γίνεται διαχωρισμό σε συγκεκριμένα θέματα, όπως συμβαίνει στην Κόζακ, αλλά γενικότερα θέματα. Ας πούμε, ε, μεταναστευτικό, προσφυγικό. Επ' αυτού να υπάρχει ad hoc κοινοβουλευτική συνεργασία για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επιληθεί το πρόβλημα. Και μέσα από την IPAX ε, μπορεί να οργανωθεί ένα φόρουμ online καταρχήν ανάμεσα στους διάφορους εθνικούς βουλευτές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ή με την κοινή γνώμη. Διότι και οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν. για μένα ένα μοντέλο, ένα πρότυπο θα μπορούσε να είναι το IGF, Intergovernance Forum, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά από πλευράς οργάνωσης ε, θα έχουμε ίσως 2.000 ανθρώπους που θα συζητάνε σε ομάδες εργασίας και ό,τι συζητάνε θα μεταδίδεται online και όποιος από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ενδιαφέρεται θα μπορεί να παρεμβαίνει και να συζητάει και αυτός online σε αυτό το δίκτυο. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών. Τελευταίο σημείο, ε, το δέκατο, οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες. Ναι, επ' αυτού. Δεν το βρίσκω κακό για να έχουμε κατά νου την Ευρώπη, αλλά σας προειδοποιώ να μην έχουμε κατά νου ότι με αυτή την, εβδομάδα τελειώσαμε με την Ευρώπη. Και για όλες τις άλλες εβδομάδες του χρόνου μπορούμε να χαράξουμε εθνική πολιτική. Αν το πιστεύουμε αυτό, αυτό είναι σε αντίφαση με αυτό που είπα στην αρχή. Ε, τα εθνικά κοινοβούλια είναι σήμερα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Δηλαδή κάθε εβδομάδα υπάρχει μια ευρωπαϊκή εβδομάδα και οι βουλευτές πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουν και να ε, καταλάβουν ότι πρέπει να ε, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη στην Ευρώπη στην καθημερινή του κοινοβουλευτική εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Καθηγητά Περνίτσε. Τώρα αρχίζουμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά στο θέμα της πράσινης κάρτας, νομίζω μετά από αυτά που είπατε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα δυνατό σημείο. Έχουμε 12 ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Όποιο θέλει να πάρει το λόγο πρέπει να συμπληρώσει αυτό το κίτρινο χαρτί, έτσι. Και αρχίζουμε. Όπως είπαμε, δύο εθνικοί βουλευτές και ένας ευρωβουλευτές. Ντανιέλ Ρουά από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που έθεσε πολλά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν εδώ και καιρό και ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες που μίλησαν εκτενέστατα σχετικά με την πράσινη κάρτα. Και εμείς ως εθνικοί βουλευτές εδώ και καιρό συζητάμε για αυτά τα θέματα και χαιρόμαστε που τα αναλύουν τώρα και οι ευρωβουλευτές. Τώρα θέλω να απαντήσω καταρχήν έτσι συνοπτικά και μετά και γραπτά θα το κάνω βέβαια, τόσο μας είπε ο συγητής. Λοιπόν, είναι σημαντικό η διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης να ληφθεί υπόψη με την αναλογικότητα. Συμπληρωματικά προς την επικουρικότητα. Δεν πρέπει το ένα να το φέρνουμε σε αντίθεση με το άλλο. Η διαβούλευση εθνικά, μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων επίσης είναι κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε αν κάνουμε την προθεσμία όχι 8 εβδομάδες, αλλά 10-12 εβδομάδες. Πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερο. Επίσης, θα ήταν καλό να επιτρέψουμε στις πολιτικές μειονότητε να εκφράζονται στις διάφορες γνωμοδοτήσει που στέλνουμε στα πλαίσια της επικουρικότητα, ώστε η άποψη των μειονοτήτων αυτών να γίνεται ε, περισσότερο κατανοητή. Επίσης, για να υποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο στα εθνικά κοινοβούλια από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να κοιτάξουμε να υπάρξει μια νέα σύγκληση στο χρονοδιάγραμμα, αλλά από την άλλη μεριά ε, η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα, τον εθνικό προπολογισμό να γίνεται πριν αρχίσει η συζήτηση επί του προπολογισμού στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί μερικές φορές ε, πέφτουν έτσι ημερομηνίε που δεν στέκει. Επίσης, για να υπάρχει θετικός ρόλος από πλευράς των Εθνικών Κοινοβουλίων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δικιά μας Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων το θέλει πάρα πολύ. Ο έλεγχος της υπηκουρικότητας είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα πρέπει, συμφωνώ, όχι με κόκκινη κάρτα να το, να χρησιμοποιούμε τη διαδικασία αυτή. Έτσι κι αλλιώς ακόμα και η κίτρινη κάρτα πιο πολύ τα διέξοδα προβάλλει παρά τα θετικά. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παίξει ρόλο γέφυρας ανάμεσα στην κοινή γνώμη και τους βουλευτές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εμείς είμαστε από τα κοινοβούλια που έχουν ήδη ε, προτείνει πράσινες κάρτες μερικές φορές. Η Κομισιόν όμως πρέπει να μας ακούει. Δεν πρέπει να λέει μα υπάρχει εδώ, υπάρχει εκεί, υπάρχει παραπέρα. Όχι. Είναι μια αντιπαράθεση που θα πρέπει συλλογικά να διαχειριζόμαστε και όχι από μόνη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, τρία ζητήματα θα έπρεπε να υπογραμμίζονται περισσότερο. Πρώτον, η εισαγωγή μιας κοινοβουλευτικής διάστασης στην Ευρωζώνη με μια διατύπωση που θα βρούμε. Έπειτα, ο διακοινοβουλευτικό διάλογος πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα για τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά ζητήματα, όπως λέει και το 13 του ΕΣΕ. Αυτό πρέπει να γίνεται και με την έγκριση συμπερασμάτων που επιτρέπεται σήμερα με εσωτερικού κανονισμούς. Και τέλος πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο. Πολυεθνικά ψηφοδέλτια θα μπορούσε να έχει νόημα Φυσικά να υπάρχει ισορροπία για τους εθνικούς εκπροσώπους που βρίσκονται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως, οι δύο ιδέες είναι ενδιαφέρουσες και θα πρέπει να τις εξετάσουμε περισσότερο. Τέλος, μια ετήσια συνάντηση, κάποιο είδους συμπόσιο, μια εβδομάδα ανάμεσα στους εθνικούς βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, θα έχει νόημα Κυρίως αν μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης. Ακριβώς αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή, πιο δημοκρατική Ευρώπη και έτσι νομίζω ότι θα μας καταλάβουν ακόμα καλύτερα και οι πολίτες μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ρετζίνα Μπάστος από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά να συγχαρώ τον εισηγητή Πάολο Ρανζέλ που είναι βαθύς γνώστης αυτών των θεμάτων και κατάφερε να προετοιμάσει ένα προκατακτικό έγγραφο τόσο καλό όσο αυτό που έχουμε σήμερα εδώ σε αυτή την πρώτη μας ε, συνεδρίαση. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η συνθήκη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια συμβάλλουν δραστήρια στην ε, εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, όπως είπε και ο πρόεδρος Καζίνη, και αυτό ε, μέσω σημαίνει ότι η ε, αναγνώριση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων και ξεπερνά, που ξεπερνά τον παραδοσιακό ρόλο του ελέγχου, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τώρα λοιπόν έχουμε αυτό το μηχανισμό πρόερες, προ, προειδοποίησης. Εμείς στη δική μας Εθνοσυνέλευση, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υιοθετήσαμε μία μεθοδολογία ελέγχου που μας επιτρέπει να απαντούμε στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις συνθήκες και έχουμε αντίστοιχα προσαρμόσει το πρόγραμμα λειτουργίας του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Ε, προχωρήσαμε λοιπόν σε μια μεταρρύθμιση της μεθοδολογίας αυτού του ελέγχου και αυτή η νέα μεθοδολογία συνεχίζει να εξελίσσεται ε, και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, στις ε, νομοθετικές συνελεύσεις των αυτόνομων περιοχών, αλλά συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών σε όλη αυτή τη διαδικασία ελέγχου. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι ο πολιτικός διάλογος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντική σημαντικό σκέλο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να είναι σαφή η αποστολή μας στο να τηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητα. Επίση, θεωρούμε πω η έκφραση της αντίθεσης της μειοψηφίας μέσω της συμπερίληψης των δηλώσεων, αιτιολογήσεων μάλλον ψήφου είναι πολύ σημαντική ε, και εδώ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια και προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα και σε αυτά τα θέματα λαμβάνοντας υπόψη και την πρόταση ε, του ίδιου του εισηγητή. Αλλά επίσης ε, ε, παρακολουθούμε μέσω μιας ιδιαίτερη, ειδικευμένης μάλλον μορφής διάφορες υποθέσεις της Ένωσης μέσω των μονίμων μας εισηγητών όπως συμβαίνει και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλα τα θέματα κοινή πολιτικής και πολιτικής άμυνας αλλά καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, με το πυλώνα που αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα αλλά και τα θέματα του Brexit τα παρακολουθούμε διαρκώς και μονίμως. Προφανώς υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν αλλά πιστεύουμε ότι με τον καιρό θα μπορέσει έτσι να δοθεί φωνή και στα εθνικά κοινοβούλια ώστε να εμβαθυνθεί ο τρόπος επαφής με την νομοθεσία που συντάσσεται εδώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά προσφέροντας μια σταθερότητα. Οι τροπολογίες που σημαίνουν μεταρρύθμιση των συνθηκών δεν θα ήταν καλό να γίνουν τώρα. Ε, ανησυχούμε, θέλουμε να ενισχύσουμε τη διακυβερνητική συνεργασία, θέλουμε να, μας, να αποκομίσουμε περισσότερα από τις συνεδριάσεις της ΚΟΖΕΚ, να εγγυηθούμε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια συνομιλούν μεταξύ τους και προσέχουν, τις δίνουν, δίνουν μάλλον βάση στις απόψεις των ΜΕΝ και των ΔΕΑ, καθώς και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετάχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψη απόφασης της Ένωσης με δυνατότητα προσφυγής στην πρωτοβουλία του, της Πράσινης Κάρτας, όπως είπε και η συνάδελφος Ντανιέλο Ρουά σε διάφορα Εθνικά Κοινοβούλια που έχουν λάβει αυτή την πρωτοβουλία του πράσινου, της πράσινης κάρτας και είμαστε και εμείς στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο μεταξύ αυτών συνέβαλε αυτό στη διαφάνεια του ελέγχου. Ε, θέλουμε να συμμετέχουμε λοιπόν πιο ενεργά στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και αναμφίβολα επίσης αυτή είναι η αποστολή που έχουμε αναλάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, εκ μέρους του σκιώδους εισηγητή και επειδή είμαι και συντονιστή, θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου δύο λεπτά και θα μιλήσω ιταλικά. Ε, το, η δική μου ερώτηση και, δικός μου, και δική μου, ο δικός μου προβληματισμός ξεκινούσε από την ερώτηση που έθεσε ο, ο εισηγητής Ρανζέλ για το θέμα της πράσινης κάρτας σε μια εκδοχή light, πιο ελαφριά, ε, μέσα σε πλαίσια δηλαδή λογικών προτάσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όμως, ή τα όσα μας, είπαν, μας είπε ο καθηγητής Περνίτση και οι υπόλοιποι που είστε υπέρ μιας ε, δυνατότητας πρότασης ε, πρωτοβουλίας και όχι δηλαδή ε, πρότασης που θα απαγορεύει ε, κάποια δράση αλλά περισσότερο μια πρόταση για εργασία. Καλό θα είναι λοιπόν να το πούμε και εμείς εδώ ως Επιτροπή Συνταγματική θα το μελετήσουμε. Θα μελετήσουμε τη δυνατότητα αυτή που ανέφερε ο καθηγητής Πέρνιτζε, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της επικουρικότητας αντίστροφα, δηλαδή να θεωρήσουμε πως είναι φυσιολογικό τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να προτείνουν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ένα θέμα που είναι ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και μπορεί να λυθεί περισσότερο, καλύτερα μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα το προτείνω στην Κομισιόν με βασιζόμενη στον έλεγχο της αρχής της επικουρικότητας η οποία μπορεί και να μην τηρηθεί, μπορεί και να μην τηρηθεί, γιατί αν δεν κάνει κανείς προτάσεις που θα μπορούσε να κάνει. Αυτό θα πρόσφερε τη δυνατότητα να μείνουμε μέσα σε μια υπόθεση πράσινης κάρτας και χωρίς τροποποίηση των συνθηκών. Διότι αυτή η δυνατότητα δίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια και αν έτσι το ερμηνεύσουμε μπορούμε να είμαστε και να μείνουμε εντός των συνθηκών χωρίς να απαιτηθεί τροποποίηση που όπως γνωρίζετε δεν πρόκειται να γίνει αύριο. Εγώ λοιπόν προσωπικά θα εργαζόμουν περισσότερο και το λέω στον εισηγητή μας για αυτό το θέμα, αλλά το προτείνω και όταν κάνετε προτάσεις να αναφέρετε την αρχή της επικουρικότητας ως μάλλον της αντίστροφης επικουρικότητας, πράγμα το οποίο είναι απόλυτα θεμητό. Και η δεύτερη παρατήρηση, που και αυτή έγινε από πολλούς, αλλά πήρε πιο τυπική μορφή στην πρόταση του καθηγητή Περνίτσε, να δούμε πώς θα έπρεπε καλύτερα να αντιποποιηθούν τα αποτελέσματα. Μήπως, όχι δηλαδή να υπάρχει ήδη αρμοδιότητα λήψης απόφασης της ΚΟΖΑ και της Επιτροπής με την, υπό το άρθρο 13, αλλά να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως προτάσεις από την Επιτροπή ή ε, να τη ζητήσει το Κοινοβούλιο μέσω του έμεσου δικαιώματος πρωτοβουλίας που έχει, τη νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι μια άλλη φάση που θα δώσει περισσότερη ισχύ στον πολιτικό διάλογο. Πρώτα θα ενισχύσει δύο εθνικά κοινοβούλια αλλά και τον πολιτικό διάλογο αυτόν που γίνεται ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Και έπειτα στη συνέχεια υπάρχει και αυτός ο διάλογος με την Κομισιόν και τα άλλα θεσμικά όργανα. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Σα ευχαριστώ και τώρα θα περάσω στην επόμενη ε, παρέμβαση. Η κυρία Μαρίνα Μπερλιγκέρη από την Ιταλία. Από το Κοινοβούλιο της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα που συζητάμε σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία στη φάση που βρισκόμαστε, δηλαδή ε, συζητάμε για τις μελλοντικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης συζητάμε και τις αλλαγές που ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων έτσι ώστε να μπορούμε και να επικαιροποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Το θέμα είναι η κοινή γνώμη και από αυτού νομίζω ότι υπήρξαν διάφορες προσεγγίσεις από διάφορες πολιτικές δυνάμεις ε, με βάση και τις εξελίξεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Σε γενικές γραμμές, οι πολίτες των χωρών μας έχουν δείξει επανειλημμένα Κυρίω κυρίως ε, με αναμφίβαλο τρόπο το ότι επιθυμούν να προσαρμοστούν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Ε, σιγά λέει η πρόεδρος. λίγο πιο αργά. Λοιπόν, ακόμα και για να ε, περιοριστεί η απόσταση που κατά την άποψη πολλών διευρύνεται συνεχώς ανάμεσα στους ε, θεσμούς για τους πολίτες και στις απαντήσεις ε, των Είναι λοιπόν σημαντικό να αξιολογήσει κανείς το ρόλο των κοινοβουλίων, τα οποία κοινοβούλια στις όριμες δημοκρατίες είναι ο βασικός χώρος όπου υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση, θεσμοθετημένη πολιτική αντιπαράθεση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αποδίδεται η μέγιστη σημασία που μπορούν να προσφέρουν τα εθνικά κοινοβούλια στην βελτίωση των ευρωπαϊκών διαδικασιών. Αυτή είναι μια δέσμευση που έχει δει προ προαγγελτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει θα δώσει μεγαλύτερη σημασία στα εθνικά κοινοβούλια κυρίως όσον αφορά τις ε, νομοθετικές πράξεις. Όμως μέχρι τώρα ε, δεν έχει υπάρξει κάτι συγκεκριμένο και μάλιστα η ε, αποφάσεις επιτροπής ε, στέλνονται με κάποια καθυστέρηση και δεν εξετάζουν τις κρίσιμες ε, παρατηρήσεις. Είναι λοιπόν προς όφελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσέχει περισσότερο σε αυτό το θέμα για να μην ε, τελικά υπάρξει ο κίνδυνος που φοβόμαστε, δηλαδή να αυξηθεί περαιτέρω ο ευρωσκεπτικισμός και η δυσπιστία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια να τα συμπεριλαμβάνει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντικές είναι και οι συζητήσεις ε, που γίνονται σε σχέση με την ε, διακοινοβουλευτική συνεργασία. Παραδείγματο χάρη, η Κόζα ε, θα πρέπει να αποφεύγει να εξετάζει πολύ γενική φύσεως θέματα, να εστιάζεται σε πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, σημαντικές πρωτοβουλίες και με τον τρόπο αυτό τα διάφορα κοινοβούλια θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και των ε, ευρωπαϊκών πολιτικών. Όχι αφηρημένα, ε, γιατί αυτά ε, συμβάλλουν να υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από τους πολίτες. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι θετική η πρόταση να, βελτιωθούν καλύτερα, να βελτιωθεί καλύτερα η συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό και να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές να συμμετέχουν σε επιτροπές και όχι μόνο στις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Εξάλλου, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερος ο έλεγχος. Και η δημοκρατική νομοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω. Με τον τρόπο αυτό το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να εκφράζει τις ε, υπερεθνικές απόψεις, κάτι που ανέφερε και ο κύριος ε, Καζίνη. Ε, αυτή λοιπόν η πρόταση περιλαμβάνεται επίσημα στο ψήφισμα που εμείς ε, καταθέσαμε στο Κοινοβούλιο μας την προηγούμενη εβδομάδα ε, μετά από τις αποφάσεις που έγιναν γνωστές από το Ευρωπαϊκό Συνοβούλιο σε σχέση με την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, Έντγκαρ Μάγερ, Αυστρία. Παρακαλώ, το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ είμαι ο Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δεύτερης Αυστριακής Βουλής. Το Bundesrat στην Αυστρία τα τελευταία χρόνια, ε, τουλάχιστον όσον αφορά την ε, επικουρικότητα έχει ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα. Μέχρι τώρα έχουμε 29 γνωμοδοτήσεις και πάνω από 40 ανακοινώσεις. Αυτές ε, αφορούν διάφορα θέματα. Δεν τολμώ βέβαια να διαφωνήσω με τον καθηγητή κύριο Περνίτσε, αλλά πρέπει να πω ότι εμείς ε, δεν είμαστε κατά της Ευρώπης, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας επικοδομητικός ε, κρίσιμος διάλογος. Ε, αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της, ε, των ευρωπαϊκών διαδικασιών. Εμείς στο Bundesrat έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τα αυστριακά κρατήδια. Το Bundesrat είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην νομοθεσία ευρωπαϊκού επίπεδου και τα κρατήδια. Αυτή λοιπόν η ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, αυτή αναγνωρίζεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την Επιτροπή των Περιφερειών. Υπάρχει το πρότυπο συνεργασίας ανάμεσα στα εθνικά ε, και τα τοπικά κοινοβούλια. Αυτό είναι ένα υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Όσον αφορά την επικουρικότητα και νομίζω αυτό το έχω ήδη πει σε συνεδριάσεις της ε, ΚΟΖΑΚ και στην ε, συνδιάσκεψη ε, της Επιτροπής των Περιφερειών για την επικουρικότητα. Είπα λοιπόν ότι εκεί πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 8 εβδομάδες. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να υπάρξει παράταση της προθεσμίας. Και όσον αφορά στη συνεργασία με τα κρατήδια, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έτσι ώστε να κλείσουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες. Εξάλλου, με τροποποίηση του κανισμού, μεριμνήσαμε να υπάρχει πιο στενός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με όλα αυτά τα μέτρα, μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη διαδικτύωση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό, το εθνικό και το τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω την κυρία Χούμπνερ και τον κύριο Ραντζέλ για το ότι οργάνωσαν τη σημερινή συνάντηση. Η συμπερίληψη των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Πολιτική, ειδικά σε μια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τόσες πολλές προκλήσεις, η συμμετοχή μας είναι εκ των όνου κάνευ. Ε, ο κύριος Ραντζέλ μας έστειλε πολλά και ενδιαφέροντα έγγραφα και αναφέρθηκε σε πολλά προφορικά. Εγώ θέλω να προσθέσω επιπλέον ένα, το θέμα των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή, η αρμόδια στο Bundesrat, έχει αποφασίσει επ' αυτού και έχει πει ότι ε, δεν αμφισβητείται η σημασία των κατεξουδότηση πράξεων. Αυτό όμως που επικρίνουμε είναι το πόσο συχνά εφαρμόζονται οι πράξεις αυτές. Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα από τη συνθήκη τη Λισαβόνας και μέχρι σήμερα έχει βελτιωθεί. Όμως η επιρροή των Εθνικών Κοινοβουλίων σε ε, κατεξοδότηση πράξης ή σε εφαρμοστικές πράξεις, τουλάχιστον κατά την άποψη του Bundesrat, δεν αρκεί και για μας θα ήταν ε, σκόπιμο το θέμα αυτό να το συζητήσουμε σε βάθος. Και τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς θα χαρούμε ιδιαίτερα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε 8 εβδομάδες μπορούσε να τοποθετείται στις γνωμοδοτήσεις μας. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Πρόεδρος, ε, πολύ καλή παρατήρηση αυτή. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Νταϊάννα Τζέιμς. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτηση και τόσα άκουσα από τους εμπειρογνώμονες βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Όλοι θυμούμαστε το βασικό πυλώνα πως είναι κανείς μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρόκειται για επιμερισμένη κυριαρχία και παρά το δημοψήφισμα και το Brexit εξακολουθούμε να είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και συμμετέχουμε. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω ένα στοιχείο κλειδί και αυτό είναι μια προσδοκία από τους πολίτες των χωρών μελών για την αποκοινού λήψη αποφάσεων. Και μια από τις μεγαλύτερες επικρίσεις που ακούγονται, κυρίως από τα ε, κόμματα κατά της Ευρώπης, είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι λαμβάνονται έτσι στα μυστικά διάφορες αποφάσεις, πράγμα που οδηγεί βέβαια σε τεράστια απογοήτευση και απομάκρυνση των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε για να το διορθώσουμε αυτό θα ήταν χρήσιμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής ε, ε, εκστρατεία ε, για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 60 με 70% των νομοθεσιών, είπαμε, απορρέουν από ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια, όμως, ακούσαμε ότι δεν ισχύει αυτό επίσης. Οπότε, αναρωτιέμαι, εδώ μιλάμε για επικουρικότητα, αλλά τελικά μήπως ε, εννοούμε ότι είναι τα εθνικά κοινοβούλια υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια σχόλια τώρα σύντομα. Αναφέρθηκε ευρωβουλευτές, εθνικοί βουλευτές, αλλάζουν καπέλο κάθε τόσο. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να το ερευνήσουμε αυτό γιατί δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρεσει με την Ολική κυβέρνηση και τη Σκοτσέζικη κυβέρνηση που εκείνοι μπορούν να έχουν διπλό ρόλο. Πολλά από τα σχόλια πάντως που άκουσα εδώ οδηγούν σε περισσότερη γραφειοκρατία κατά τη γνώμη μου και κάνω έκκληση στον κόσμο. Αυτό είναι που πρέπει να ε, διώξουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη γραφειοκρατία δεν είναι δυνατό να συνεχίζεται αυτή η τάση της γραφειοκρατίας. Δεν είναι δυνατό να ζητάμε να γίνονται συζητήσεις και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και να σας πω ακόμα είναι δυνατό να ζητάμε τώρα να μπει άλλο ένα στρώμα, άλλο ένα επίπεδο. Έχουμε τη Βουλή των Λόρδων, τη Βουλή των Κοινοτήτων στον Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς ζητάτε ένα τρίτο στρώμα. θα έπρεπε όλες οι χώρες μέλη να προσπαθούν να απλοποιήσουν τα πράγματα και να έχουν περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες, όχι το αντίθετο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ιωάννης Σαρακιώτης τώρα έχει το λόγο από τη Βουλή των Ελλήνων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους προλαλήσαντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια κρίσιμη περίοδο καθώς καλείται να δώσει πιστικές απαντήσεις σε μια σειρά από προκλήσεις από την παγκοσμιοποίηση και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία, την απασχόληση μέχρι την ασφάλεια, την προσφυγική κρίση και την άνοδο του λαϊκισμού ανταποκρινόμενη πάντοτε στις ε, απαιτήσει των πολιτών η Επιτροπή Γιούνκερ ανέλαβε κάποιε πρωτοβουλίε για τη βελτίωση του συντονισμού των οργάνων τη, όπω για παράδειγμα την αναθεώρηση τη διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθέτηση. Είναι γεγονό ότι ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, σύμφωνα με τη συνθήκη, συνίσταται κατά βάση στη μέρημνα τη στήριση τη αρχή τη επικουρικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμω, ανεξαρτήτως του θεσμικού ρόλου που προβλέπει η συνθήκη στα Εθνικά Κοινοβούλια, πολιτικά είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί ο ουσιαστικός τους ρόλος, καθώς αυτά αποτελούν και τον εγκύτερο προς τους πολίτες δημοκρατικό θεσμό, με τους εκπροσώπους τους να έρχονται σε καθημερινή επαφή με την κοινωνία των πολιτών και να αποτελούν το βασικό συνδετικό κρίκο με τα κέντρα λήψης αποφάσεων θα μου επιτρέψετε με την ευκαιρία και καθώς συζητούμε μεταξύ άλλων για τα όρια των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων να κάνω μια ειδικότερη παρατήρηση. Είναι γεγονός ότι ορθώς γίνεται μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσης της γραφειοκρατίας και συντόμευσης των νομοθετικών διαδικασιών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει με αυτή τη δικαιολογία να γίνεται καταχρηστική χρήση των διατάξεων της συνθήκης. Συγκεκριμένα σημειώνεται τάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επικαλείται τις διατάξεις 290 και 291 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύω με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών. Η χρήση των εν λόγω άρθρων θα πρέπει να γίνεται με φιδό ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτική ώστε να μην υπερβαίνει τις εξουσίες της σε σχέση με την έκταση της εξουσιοδότησης. Προσφάτως, η Βουλή των Ελλήνων εξέδωσε γνώμη επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και, επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά. Στην αιτιολογική έκθεση της νέας πρότασης υπογραμμίζεται ότι αυτή εισάγει μόνο μερικές ίσονος μικρότερης σημασίας τεχνικές τροποποιήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή του προηγούμενου κανονισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εισάγει αριθμό κατεξιοδότηση πράξεων. Στην πραγματικότητα όμως οι πράξεις αυτές εισάγουν και νέα ουσιώδη στοιχεία στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 290. Κάνω λοιπόν έκκληση στην Επιτροπή να επανεξετάσει τον εν λόγω κανονισμό, καθώς επίσης και να είναι πιο προσεκτική στην εφαρμογή των άρθρων 290 και 291. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. είναι ο κύριος Βιταλίνο Κάνας από την Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή πρόεδρος μάλλον τη Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου σας έδωσε μια ε, ζωηρή εικόνα για την καθημερινότητά μας και το πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο μας ε, για να συγχαρώ τον επισηγητή ε, Παύλο Χανζέλ που μα έδωσε τόσο πολύ εμπεριστατωμένη έκθεση και θα αρχίσω με μια ενοιολογική σημείωση που είναι η εξή. Τα εθνικά κοινοβούλια, τα δημοκρατικά κοινοβούλια εν γέννη, ε, έχουν ε, ε, ένα σύνολο βασικών ιδεών επί των οποίων στηρίζονται. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν εκλήγονται, δεν έχουν δημοκρατική νομιμότητα για να δίνουν γνωμοδοτήσεις, να αναλάμβουν πρωτοβουλίες ή να στηρίξουν τέτοιες πρωτοβουλίες κτλ. Όμως αυτοί οι μηχανισμοί που περιλαμβάνονται στο συνθήκη της Λισαβόνας στο 12ο άρθρο είναι μηχανισμοί πολύ σημαντικοί ώστε τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι περιορισμένοι ε, ε, περιορισμένου εύρους ε, μέσα, αυτό η κίτρινη κάρτα, η πράσινη κάρτα κτλ. δεν συμβαδίζουν με την καθημερινή δημοκρατική ζωή των κοινοβουλίων επιπλέον. Αυτά τα μέσα, τα τεχνικά και τα νομικά πολύ δύσκολα τα χειρίζονται οι πολιτικοί των εθνικών κοινοβουλίων γιατί η αρχή της επικορικότητας έχει πολιτική διάσταση αλλά πάνω απ' όλα έχει και τεχνική και νομική διάσταση. Τα εθνικά κοινοβούλια πολύ συχνά δεν δυσκολεύονται να το χειριστούν το ίδιο και για την αναλογικότητα. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως τα εθνικά κοινοβούλια θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να ευαληθεύουν κατά πόσο τηρείται η αρχή της αναλογικότητας αλλά και, είναι, και αυτή η αρχή τόσο δύσκολη από τεχνική και οικονομική άποψη που είναι πολύ ε, ε, δυσχερές να τον ελέγξουν τα εθνικά κοινοβούλια. Τούτου λεχθέντος τι πιστεύουμε ότι περιμένουν οι πολίτες μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλουν να ασκήσουν τις, τα καθήκοντα για τα οποία εξελέγησαν, δηλαδή έλεγχος του εκτελεστικού και, της και πρόταση της νομοθεσίας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε μέσα σε αυτή τη μελλοντική μας προοπτική να αναζητήσουμε τους μηχανισμούς που θα συμμορφωθούν με την διολογική αυτή δημοκρατία των κοινοβουλίων γίνει λόγος για την κόκκινη κάρτα και διαφορετικές απόψεις για την κόκκινη κάρτα. Εγώ θα ήμουν προσωπικά υπέρ της κόκκινης κάρτας γιατί ε, ήδη η κίτρινη κάρτα θα χρησιμοποιείται λίγο αλλά η κόκκινη ακόμη πιο λίγο. Όμως ε, σημαίνει μια απόδοση πραγματικής αρμοδιότητας στα, ευρωπαϊκά, στα εθνικά κοινοβούλια που θα μπορούσαν όντως να καθορίσουν, να υποχρεωθούν να αναλάβουν κάποιες πρωτευουλίες. Όχι αναγκαστικά να χρησιμοποιήσουν την κόκκινη κάρτα αλλά να αναγκαστικά να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες, να παρακολουθούν και να εξετάζουν τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες <coughs> και θα είχαν μια πιο πραγματική έτσι, αρμοδιότητα. Δέχομαι ωστόσο πως ε, το, η κόκκινη κάρτα περιλαμβάνει και αρνητικά στοιχεία για τις οποίες θα έπρεπε να αναθεωρηθεί η συνθήκη αν θέλαμε να τις διορθώσουμε και όλοι είμαστε κατά αναθεώρηση συνθήκης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάποια μέσα για τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να μπορέσουν να δουν τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει κάθε φορά. Και εγώ θα έλεγα λοιπόν κίτρινη κάρτα αυτήν που πρότεινε ο Παύλο Ρανζέλ και την πράσινη κάρτα. Ήδη είπαμε ότι εμείς αυτό προωθούμε στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε πως είναι μια ενδιαφέρουσα ε, πρόταση, αν και περιορισμένη, γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί διευρυμένη συνένεση ανάμεσα σε διάφορους ε, πρωτοβουλευτές, ώστε να είναι ισχυρές οι πρωτοβουλίες που προκύπτουν την πράσινη κάρτα, αλλά ε, αυτή η πρόταση η οποία είναι πολύ καλή είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Ίσως όχι ακριβώς όπως το είπατε, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κάθε χρόνο η Κομισιόν παρουσιάζει το δικό της ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν μία τέτοια ε, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ε, πριν η Κομισιόν να παρουσιάσει το δικό της πρόγραμμα εργασίας ε, ώστε τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να ε, ελέγξουν, να εξετάσουν ένα πρόγραμμα, σχέδιο προγράμματος εργασίας της Κομισιόν για να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια, να ελέγξουν το εκτελεστικό ε, και σε αυτή την περίπτωση να ελέγξουν το εκτελεστικό την Κομισιόν, την εκτελεστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ καλή πρόταση λοιπόν του Πάολο Ροζέλ να δούμε πώς, ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την εφαρμογή της χωρίς να αναθεωρηθεί η συνθήκη συμφωνούμε. Θεωρώ όμως ότι αυτό θα επέτρεπε να κινητοποιηθούν οι εθνικοί βουλευτές για πιο ε, προσεκτική εργασία για τα ευρωπαϊκά θέματα και μεγαλύτερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά θέματα. Ευχαριστώ. να. Ραμόν Αουρέγγι. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που ήρθαν εδώ σήμερα. Αυτούς που ήρθαν κυρίως, έτσι. Γιατί πολλές χώρες δεν έστειλαν εκπροσώπους, κάτι το οποίο είναι πολύ κρίμα κατά τη γνώμη μου. Και ευχαριστώ και τον κύριο Ρανζέλ και όλους τους εμπειρογνώμονες που μας προτείνουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος για να είμαστε και ξεκάθαρη για τις απόψεις μας. Πρώτον, έχω την αίσθηση ότι η έκθεση για την επικουρικότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων εν μέρη εξαιτία αυτών που είπαν εδώ ότι πρόκειται για μια ε, νομική τεχνική πολύ περίπλοκη, τελικά έχουν καταλήξει να γίνονται μια τεχνική φύσεως ρουτίνα. Εγώ ήμουν βουλευτή στη χώρα μου και θυμάμαι ότι συμμετείχα στις εκθέσεις αυτές για την επικουρικότητα και τα πολιτικά κόμματα στη χώρα μου, στην Ισπανία, ειλικρινά δεν δούλευαν πάνω στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δηλαδή μα ζητούσαν να διαβάσουμε την έκθεση των νομικών εμπειρογνωμόνων και αν εκείνοι έλεγαν δεν υπάρχει πρόβλημα, Λέγαμε κι εμείς, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν όμως ότι η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να εμπλουτιστεί. Έγιναν κάποιες προτάσεις εδώ. Και κυρίως λαμβάνοντα υπόψη ότι στην Ευρώπη έχουμε πολλές χώρες μέλη που διαθέτουν ένα σύστημα περιφερειών όπου υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων στις αυτόνομες περιφέρειες, στην Ισπανία, στα Λέντα, στη Γερμανία κλπ. Άρα πρέπει η έκθεση να συμπληρωθεί και με τη συνεισφορά των ε, Λέντερ, για παράδειγμα, όπως μας είπε ο Αυστριακός συνάδελφος, και από τις μειονότητες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να γίνει για να εμπλουτιστεί η αρχή της επικουρικότητας. Δεύτερον, πράσινη κάρτα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα, γιατί δίνει την ευκαιρία σε συνεργασία για διάφορες πρωτοβουλίες. και για την κίτρινη κάρτα. Εντάξει, αλλά είμαι εντελώ κατά τη κόκκινη κάρτα. Δεν θέλω τώρα να επαναλάβω τα επιχειρήματα που είπαν πολλοί συνάδελφοι εδώ ήδη πριν από μένα. Αυτό όμω που έχει σημασία κατά τη δικιά μου γνώμη είναι τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν ένα επίπεδο συζήτηση για την Ευρώπη που να γίνεται πιο συχνά και με πιο έντονη απόχρωση. Ο έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων έλεγχος των επικεφαλής των κυβερνήσεων που πηγαίνουν στο Συμβούλιο ή τους εκπροσώπους που πηγαίνουν στο Συμβούλιο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ και 8 χρόνια είμαστε σε οικονομική κρίση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο κατέληξε να είναι ένα όργανο με υπερβολικά μεγάλη δύναμη σε σχέση με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο δηλαδή αποκτά όλο και περισσότερε εξουσίε και αρμοδιότητε και παίρνει αποφάσει που έχουν να κάνουν με του πολίτε, τη διακυβέρνηση τη ε, κρίση για παράδειγμα. Οπότε το ζήτημα είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συζητάνε τις αποφάσεις που παίρνουν αυτοί που τους κυβερνούν και που τις παίρνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια που είναι στην Ευρώπη να συζητούν για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο Πάολο Ρανζέλ μας πρότεινε διάφορους μηχανισμούς. Εμένα μου κάνουν όλοι. Και θα πρότεινα και κάτι ακόμα. Μία παρουσία, δεν θα έλεγα μία εβδομάδα το χρόνο, αλλά στις μεγάλες συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ή για διάφορες κρίσεις, όπως η οικονομική κρίση, προτείνω να έχουμε συζητήσεις στα εθνικά κοινοβούλια και με τους ευρωβουλευτές της λόγω χώρας και με επιτρόπους. Γιατί είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα εθνικά κοινοβούλια. Πάντα βέβαια σεβόμενοι τις αρμοδιότητες του καθενός, έτσι. Και συγχρόνως να υπάρχει και μεγαλύτερη συνεργασία μέσα στα εθνικά κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στα πλαίσια μιας ε, εξεταστικής επιτροπής. Εμείς εδώ έχουμε εξεταστικές επιτροπές, κάναμε για την Ευρωπαϊκή Φορολογία, για τα Panama Papers, για τις εκπομπές οχημάτων και τους ρήπους των οχημάτων. Εδώ χρειάζεται κάποιος χώρος συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί, γιατί τελικά όλοι έχουμε τη θέση μας είτε τα Εθνικά Κοινοβούλια είτε τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών μας. Όταν πρόκειται λοιπόν για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν 500 εκατομμύρια πολίτες, ε, καταλαβαίνετε ότι για αυτούς πρέπει να δουλεύουμε. Άρα αυτή η συνεργασία είναι αναγκαία ανάμεσα στους δύο. Αυτό που λείπει σήμερα είναι να μιλούν περισσότερο για την Ευρώπη τα εθνικά κοινοβούλια και να μην θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά ζητήματα βρίσκονται στο περιθώριο των δραστηριοτήτων τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ραμόν, η κυρία Καταλίν Σόμπορ. Ουγγαρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αλήθεια, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Οι δύο παρατηρήσεις μας. Σύμφωνα με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας, υπάρχει ρόλος για τα εθνικά κοινοβούλια στην ευρωπαϊκή διαδικασία και αποκτώ και μεγαλύτερη σημασία. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο τον ρόλο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις λοιπόν των εθνικών βουλευτών. Όμως, πώς θα γίνει αυτό στο νομοθετικό τομέα, γιατί υπάρχει μία διαδικασία τριμερούς διαλόγου. Κάτι που είναι αποφασιστική σημασία στις Βρυξέλλες, αλλά που είναι άγνωστο στο ευρύ Σύμφωνα με τις έρευνες, περίπου 40% των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εξεταστεί σε τριμερή διάλογο, δηλαδή σε πέντε που γίνονται κάθε εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά τριμερής διάλογος δεν έχει νομική υπόσταση και δεν εμφανίζεται στις συνθήκες. Ούτε το κοινό, ούτε τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τρόπο για να ενημερωθούν για τις συζητήσεις που γίνονται εκεί. Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά για να επιταχυθούν οι διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, δεν υπάρχει όμως διαφάνεια σε αυτούς, ούτε δημοκρατία. Η διαδικασία των τριμερών διαλόγων λαμβάνει η χώρα στα κρυφά με την συμμετοχή των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αγαπητοί συναδελφοί, θέλω εδώ να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν καμία δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. Ο τριμερής διάλογος είναι μια διαδικασία που τίνει να γενικευθεί και είναι μια πρακτική που αποδυναμώνει το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, ο οποίος προβλέπεται αυτός στη συνθήκη της Λισαβόνας. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το τόσο σοβαρό φαινόμενο. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να περιοριστούν οι τριμερείς διάλογοι. Τότε θα λειτουργούσε καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενος. είπε η Περβάν Μπερές, Ευρωβουλευτής. Παρακαλώ. Και σκιώδησε εισηγήτρια από τους σοσιαλιστές για την έκθεση του συναδέρφου Ράνζελ. Ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή αυτή που έχετε προβλέψει σήμερα. Πρέπει να έχουμε περισσότερες τέτοιες συναντήσεις όσο μάλιστα περισσότερο ε, τα θέματα που εξετάζουμε είναι θέματα και εθνικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής ε, ε, κυριαρχίας. Και με κάποια νοσταλγία, αλλά είναι και επίκαιρο το θέμα, πολλές φορές αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Βδομάδα και είναι μια πρόταση το να δημιουργηθεί δηλαδή κάτι που να το ονομάζουμε κογκρέσο, που όμως θα έπρεπε, αν υπάρξει, να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, να καταφέρουμε όλοι να συμφωνήσουμε για το πώς, πότε θα γίνεται. Γιατί είναι όλο και περισσότερα τα θέματα πάνω στο οποία έχουμε επιμερισμένη αρμοδιότητα και κυριαρχία και είναι δύσκολο μερικές φορές να ξεχωρίσουμε τις αρμοδιότητες του μεν και, των μεν και των δε. Όσο, και, όσο περισσότερα πράγματα ακούμε, λοιπόν, για το τι γίνεται εκ παραλλήλου ε, στις 27 χώρες για το Brexit για παράδειγμα βλέπουμε ότι υπάρχει μια απομόνωση. Το Brexit όμως θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για να διορθώσουμε την ε, λειτουργία μας. Και κατά κάποιο τρόπο τελικά το Brexit μας αναγκάζει να εξετάσουμε το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα εθνικά κοινοβούλια για ένα αποτέλεσμα που σίγουρα είναι περίπλοκο. Δεν λέω ότι φταίνε οι εθνικοί βουλευτέ για τον Brexit, έτσι, μην με παρεξηγήσετε, δεν είναι αυτό που λέω. Αλλά λέω ότι αν οι εθνικοί βουλευτέ συμμετείχαν περισσότερο στα ευρωπαϊκά ζητήματα, ίσως θα μπορούσαν και καλύτερα να αντιμετωπίσουν αυτούς οι οποίοι εκφράζονταν υπέρ του Brexit. Στο Ενωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έτσι, αλλά και όχι μόνο. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, οι Βρετανοί αποφάσισαν όπως αποφάσισαν. Θέλω να έρθω τώρα σε τρία επιπλέον στοιχεία. Πρώτον, βλέπω ότι ανοίγει και πάλι η συζήτηση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Ωραία, να χρησιμοποιούμε όλες τις έννοιες, αλλά εμένα αυτό που με νοιάζει είναι το αποτέλεσμα. Ο Φιλίπ Σέγγεν ήταν ε, ένας ε, της Γαλλίας υπέρ ε, του κράτους της Γαλλίας και είχαμε τον Κλαουσιάνς που ήταν σοσιαλιστής γερμανός φεντεραλιστής και διαφωνούσαν για αυτό το θέμα. Γιατί τελικά όντω την επικουρικότητα άλλοι τη βλέπουν σαν έναν τρόπο να ανακτήσουν την κυριαρχία και άλλοι τη βλέπουν σαν έναν τρόπο να επιμεριστούν την κυριαρχία. Το ίδιο ισχύει και για την αναλογικότητα. Η αναλογικότητα χρησιμοποιείται μερικέ φορέ για να ξεφύγουμε από το γενικό κανόνα. Δεν είναι όμω έτσι που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την αναλογικότητα. Οπότε σε αυτή τη συζήτηση οριμάζει η ιδέα της πράσινης κάρτας και χαίρομαι. Όχι για να αντικαταστήσει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας που έτσι καλλιώς δεν υπάρχει, αλλά για να αρχίσει μια δουλειά σε αρμονία με τα όσα επιθυμούν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι το εξή: πάντα στα πλαίσια του Brexit ή της ευάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, Αυτά είναι θέματα τα οποία σίγουρα θα είναι πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη. Αλλά σήμερα το απόγευμα δεν συζητάμε περισσότερο για το τι σημαίνει αυτό. Εγώ είμαι κατά, το λέω εξ αρχή, ενό κοινοβουλίου τη Ευρωζώνη, όπου θα συμμετείχαν μόνο εθνικέ βουλευτέ. Δεν έχω χρόνο τώρα να το αναπτύξω περισσότερο, αλλά το κάθε κοινοβουλευτικό επίπεδο συμμετέχει στην διακυβέρνηση. Αυτό πρέπει να γίνεται όντω και πρέπει να το συζητήσουμε παρετέρω. Τέλος, το θέμα τώρα των ε, ε ψηφοδελτίων από πολλές χώρες. Το έχουμε ξανασυζητήσει και έχουμε έναν από τους συνεισηγητές. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να καταργήσουν όλες τις έδρες που κατέχει σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν όλα να μεταφερθούν σε εθνικά ψηφοδέλτια όλε αυτέ οι θέσει και αυτοί που θέλουν να βρουν μια μέση οδό. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη τελευταία λύση για πολλού και διάφορου λόγου. Πρώτα απ' όλα, γιατί από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία στην εκπροσώπηση των χωρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι αρνητικό. Μόλις στεγνώσει το μελάνι βέβαια τη συνθήκη, είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί αυτή η ανισορροπία, γιατί της καλλιώς η απόφαση παίρνεται ομόφωνα στο Συμβούλιο. Ένας από τους τρόπους λοιπόν να συμφωνήσει το Συμβούλιο για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των εθνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα, μια ποσόστοση των Βρετανικών εδρών, ώστε να υπάρξει αυτή η επανισορρόπηση στην εκπροσώπηση των χωρών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατά τη γνώμη μου αυτό επήγει να γίνει. Γιατί αν δεν υπάρξει δημοκρατική εκπροσώπηση έχουμε πρόβλημα. Τι να πούμε λοιπόν τώρα για αυτά τα ψηφοδέλτια, τα πολυεθνικά. Εγώ εδώ και πολύ καιρό έχω εκλεγεί και κάνω εκστρατεία υπέρ ενό τέτοιου ψηφοδελτίου. Στην τελευταία θητεία δεν το συζητήσαμε καν, δεν μπορέσαμε. Οπότε εγώ συμφωνώ να συνεχίσουμε να προωθούμε την πρόταση αυτή, αλλά δεν θα ήθελα να φέρει σε αδιέξοδο το σύνολο της πρότασης. Το Κοινοβούλιο θα κάνει μια νομοθετική πρόταση, ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εράρχηση στις προτεραιότητές μας. Η προτεραιότητα είναι να υπάρξει καλύτερη ισορροπία και δίκαια ισορροπία μεταξύ των χωρών μελών στην εκπροσώπησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Είμαστε από τις χώρες που έπρεπε να έχει ε, κάποιες, δηλαδή έπρεπε να έχουν δύο θέσεις λιγότερες και κάποιες άλλες όπως η δικιά μου θα έπρεπε να έχει και 11 παραπάνω βουλευτές. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει και πρέπει να συζητηθεί. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Αν τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο για, μια πολυ... για ένα πολυεθνικό ψηφοδέλτιο, φυσικά και θα ήμουν υπέρ. Αλλά δεν θα πρέπει το ένα να αποτελέσει προϋπόθεση για το άλλο, γιατί τότε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Έχουμε άλλους δύο. Κασιμίρα Ζοντόσκι, Ευρωβουλευτής. Παρακαλώ. Pani Σανόβνη ε, ε, και κύριοι, πιστεύω ότι είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το να αναζητήσει τον ε, ειλικρινή πολιτικό διάλογο ε, με τα εθνικά κοινοβούλια. Ως εκ τούτου πρέπει να διαφωνήσω με τον κύριο Περνίτσε σε δύο θέματα, κυρίως όσον αφορά στα ευρωπαϊκά θέματα που συζητούνται σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι το δημοψήφισμα που οδήγησε ε, στην έξοδο της Μεγάλης οι εκλογές στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Όλα αυτά δείχνουν ότι εστιάζουμε σε ευρωπαϊκά θέματα και νομίζω ότι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων για να βγούμε από την κρίση θα ενισχυθεί περαιτέρω. Ως εκ τούτου πρέπει να εστιάσουμε στον ε, εθνικό διάλογο, στον διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβουλία. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητάει με τις ε, μειονότητες ε, κάποιων κοινοβουλίων και αυτός είναι ένας από τους τρόπους για να οργανώσουμε καλύτερα την πολιτική μας ζωή. Και αυτό είναι αντίθετο με την εντολή που έχουν λάβει οι βουλευτές διότι οι βουλευτές, ε, οι εθνικοί βουλευτές έχουν την εντολή να ασχολούνται με νομοθετικά θέματα και όχι με αυτά που συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Εκτό, βέβαια του ότι εκπροσωπούν τα κοινοβούλια τους σε κάποια φόρουμ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε πολύ από το στόχο μας. Και τώρα όλη αυτή η συζήτηση για την πράσινη και την κόκκινη κάρτα. Ξέρετε, αυτό το εργαλείο σε κάποιο βαθμό δεν είναι λογικό. Δεν θα ήταν λογικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει να τοποθετηθεί θετικά στα σπάνια παραδείγματα της ε, κίτρινης κάρτας ε, Όλο αυτό ακολούθησε τελείως διαφορετικό δρόμο. Νομίζω η ιδέα της ε, κόκκινης κάρτας ε, προκύπτει από το γεγονός ότι αγνοήθηκε η κίτρινη κάρτα. Εγώ ε, συμφωνώ με την ανάλυση που παρουσίασε ο κύριος Ντόρν. Νομίζω ότι η αρχή της επικουρικότητας είναι η αρχή του είτε ναι είτε όχι. όπως ε, και με τον ο κύριος Χάμπλ και ο κύριος Ντόρν και εγώ θα ήθελα να υπάρχει στο μέλλον ε, περισσότερος ε, πολιτικός διάλογος που ακόμα δεν έχει όμως παγιωθεί στις συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δείξουν πόσο στενά είναι συνδεμένα μεταξύ του τα δύο αυτά όργανα για να ε, διεξάγουν ένα ειλικρινή διάλογο. Αυτά ε, είχα να πω προς τον κύριο Ρανχέλ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που οργάνωσε την ακρόαση και δούλεψε πάνω στο κείμενο που μας κατέθεσε. Ίσως λοιπόν κύριε Ρανχέλ θα άξιζε τον κόπο να παρουσιάσετε κάποιους ε, μηχανισμούς που μπορούν να συσταθούν για να υπάρχει αμυγής ε, πολιτικός διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια με θέμα την αρχή της ε, αναλογικότητας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ε, θα ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα χαρακτήριζαν αυτήν την έκθεση. Πρόεδρος, τελειώσαμε. Δεν έχω άλλους ομιλητές για πέντε λεπτά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στους εμπειρογνώμονες και μετά στον κύριο Ραγχέλ. Ο κύριος Ντόρνο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τόσο στην έκθεση του κυρίου Χανζέλ, όσο και στη διάρκεια της συζήτησης, προχωρήσαμε στην ε, κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Πιστεύω πως αυτό το καταφέραμε, μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Η απόψινή συζήτηση στην ουσία μας οδήγησε σε δύο σύνολα προτάσεων. Το πρώτο σύνολο συστάσεων θα το όριζα ως συστάσεις ε, για την εμβάθυνση στο όσα γίνονταν μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε εθνικά ε, κοινοβούλια τα οποία κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται μακριά, είναι απομακρυσμένα, αλλά θα είχαμε δηλαδή μία οργάνωση από πλευράς του ε, Κοινοβουλίου της εσωτερικής ε, ζωής της, ε, και της πολιτικής των Εθνικών Κοινοβουλίων. Βέβαια, το πρόβλημα για κάτι τέτοιο θα ήταν τεράστιες αντιστάσεις για μια τέτοια ιδέα και μάλιστα δεν θα εξυπηρετήσουν αυτόν τον ευγενή σκοπό Ιδιαίτερα να σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη ε, ε, ε, κατάσταση λόγω της κρίσης. Το δεύτερο σύνολο όμως των προτάσεων στις οποίες αισθάνομαι να είμαι πιο κοντά αναφέρεται σε αυτό που ο Στράους ονόμαζε κατασκευή από τα κάτω προς τα πάνω αλλά με πολύ στερεό και συμπαγή τρόπο. Δηλαδή πιο, κάτι, κάτι πιο ε, ε, περιορισμένο, κάτι πιο ταπεινό και σεμνό, αλλά ε, που είναι πολύ πιο στέρεο και συμπαγές. Όχι δηλαδή γοτικού τύπου οικοδομήματα τεράστια. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ο εισηγητής, δηλαδή μιλά για την αρχή της επικουρικότητας, αλλά ταυτόχρονα μιλά για το πώς θα μπορέσουμε εμείς να αναλάβουμε κάποιες από αυτές τις προτάσεις που αναφέρονται στην πράσινη κάρτα. Βέβαια δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι θα προκύψει, αλλά θα πρέπει ούτως ή άλλως να πειραματιστούμε ε, κάπως, ε, γιατί κατά τα λοιπά είμαστε αρκετά σίγουροι. Δεν είναι σίγουρο το τι θα προκύψει, αλλά σίγουρα δεν θα καταστραφεί τίποτα εάν ε, ε, προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή την ξεκάθαρη ιδέα. Θα πρέπει δηλαδή να δουλέψουμε χωρίς να θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα και χωρίς να θέλουμε να καταστρέψουμε οτιδήποτε. Ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε στη συζήτηση και τον εισηγητή. Ευχαριστώ και τώρα ο καθηγητής Περνίτσε. εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες αυτές τις συζητήσεις, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Και είμαι σίγουρη ότι έμαθα περισσότερα από αυτά που μπόρεσα να συνεισφέρω. Τρεις ε, σύντομες παρατηρήσεις θα μου επιτρέψετε. Η πρώτη μου αφορά τον εκπρόσωπο του Bundesrat της Αυστρίας. Ξέρετε, εγώ ε, παρακολουθώ τη Γερμανία, το γερμανικό σκηνικό ε, και στη Γερμανία υπάρχει αυτή η αμυντική στάση έναντι της Ευρώπης. Γι' αυτό η Αυστρία, αν έχει αυτή την επικοδομητική στάση, πραγματικά σας συγχαίρω. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο αφορά το θέμα της ε, επικουρικότητας ε, σε σχέση με τον έλεγχο των αρμοδιοτήτων και της ε, αναλογικότητας. Η δική μου εντύπωση για την εξήγηση γιατί η επικουρικότητα εντάσσεται στο σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης αλλά όχι με απόλυτη σαφήνεια. Ο λόγος ε, θα μπορούσε να είναι ότι όσον αφορά τις αρμοδιότητες, ε, το συνταγματικό δικαστήριο είναι εκείνο που αποφασίζει. Βεβαίως, ε, τίθεται το θέμα των αρμοδιοτήτων, αλλά η πεμπτουσία, το κατά πόσον υπάρχουν αρμοδιότητες ή όχι, αυτό είναι ένα νομικής φύσεως θέμα και πρέπει να παραμείνει τέτοιο, έτσι ώστε και να υπάρχει και η τελευταία σαφής απόφαση το ίδιο και για την αναλογικότητα και από αυτού υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, νομικές απόψεις ε, για το πώς ορίζεται η αναλογικότητα. Αυτό όμως δεν ισχύει για την επικουρικότητα, γιατί η επικουρικότητα είναι ένα καθαρά πολιτικό θέμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν θα αποφασίσουμε να επεκτείνουμε τα κριτήρια στο σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτά πάντα κανείς θα τα έχει κατά νου όταν μιλάει για την οπικουρικότητα, αλλά θα πρέπει ίσως ε, να διαφυλάξουμε την, τον διαχωρισμό. Κάτι άλλο που αφορά ε, στην ε, διοκοινοβουλευτική συνεργασία που συνδυάζεται με το σύστημα της πράσινης κάρτας. Εγώ καταλήγω στο ότι τελικά θα πρέπει να έχουμε διακοινωτικό διάλογο με στόχευση. Δηλαδή ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια. Στοχευμένες συζητήσει σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Είτε προτάσεις της Κομισιόν, ας πούμε, για την προστασία των δεδομένων, είτε για έναν τομέα που ακόμα δεν έχει επιληθεί, όπως είναι η πολιτική για τους πρόσφυγες. Ή TTIP, ή SETA στο παρελθόν τέτοιου είδους ε, θέματα στον, ε, να συζητούνται σε διακοινοβουλευτικό διάλογο και να εκμεταλλευτούμε αυτό το φόρουμ έτσι ώστε να καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση για την πράσινη κάρτα, μια πρόταση που θα στηρίζεται από πολλούς βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού θα έχει γίνει ε, ψηφοφορία ε, μετά αυτή η πρόταση να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό κατά την άποψή μου θα βοηθούσε πολύ και θα είχε και μεγάλη επιτυχία αν ε, ήταν και λογική βέβαια η πρόταση, πράγμα που σαφώς και το ε, περιμένω από τα κοινοβούλια. Στην περίπτωση αυτή, μια τέτοια πράσινη κάρτα θα βοηθούσε πάρα πολύ και ίσως ε, το Κοινοβούλιο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φόρουμ για την ε, επικουρικότητα σε σχέση με την έγκαιρη προειδοποίηση. Αν ε, οι βουλευτές συμφωνήσουν επ' αυτού, τότε πράγματι μπορούν να τοποθετηθούν και για την έγκαιρη προειδοποίηση. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να είμαι εδώ και να σκεφτώ κι εγώ μαζί σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ τους εμπειρογνώμονες για τα συμπεράσματα και τις απαντήσεις ο Παόλο Ραντζέλ, ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Για να δούμε αν μπορώ να συνοψίσω τις ιδέες μου. Θα αρχίσω με το θέμα της κόκκινης κάρτας. Συμφωνώ με τον γερουσιαστή Χάμπλ και με πολλούς άλλους που παρενέβησαν. Η δυνατότητα χρήσης της κόκκινης κάρτας, και εδώ έρχομαι στο σεβασμό με τον καθηγητή Περνίτσε, είναι ότι αν χρειάζεται κάτι που να μην φτάνει η κίτρινη ή η πορτοκαλιά κάρτα, τότε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για την κόκκινη κάρτα. Αλλά τότε χρειάζεται αλλαγή στην συνθήκη, οπότε είναι τεχνητό το ζήτημα. Αντίθετα, η πράσινη κάρτα όμως, που στηρίζω απόλυτα και βλέπω ότι είναι γενικά αποδεκτή, θα μπορούσε να διευκολυνθεί. Η χρήση της δηλαδή. Θα μπορούσαμε για την πράσινη κάρτα να έχουμε ως προϋπόθεση να μην ε, υπάρχουν τόσα απαιτήσει όπως υπήρχαν πριν για την κίτρινη κάρτα. Αλλά από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ για αυτό το θέμα, φάνηκε ότι κάποιοι έχουν πολύ έξυπνες παρατηρήσεις, ότι μια πράσινη κάρτα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τελικά σαν κόκκινη κάρτα. Γιατί αν έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία και κάποιος κάνει πρόταση να αποσυρθεί η νομοθεσία αυτή, τότε έχετε την προϋπόθεση να κάνετε αυτή τη συζήτηση. Είναι βέβαια μία πρόταση. Οπότε δεν νομίζω να είναι πραγματικά πρόβλημα αυτό. Και γι' αυτό και διαφωνώ με τους Πορτογάλους συναδέρφους και την Ρίτα Μολικάνες που είναι νομικός και που λέει ότι επικεντρωνόμαστε σε κάποιες εξουσίες που δεν είναι και το κέντρο των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πω όμως κάτι που υπογράμμισε και κάποιος άλλος και που στηρίζω απόλυτα, ότι δηλαδή το βασικό της αρμοδιότητας των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπετε ότι κάποια εθνικά κοινοβούλια στις κατηναδικές χώρες, για παράδειγμα, το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Και όχι μόνο στο Συμβούλιο Υπουργών, αλλά ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι έτσι κάπως ιδιόρυθμο πολιτικό όργανο γιατί συμμετέχουν οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων που εκφράζουν τις πολιτικές γραμμές της Ένωσης. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική δουλειά των κοινοβουλίων, ο έλεγχος. Από την εμπειρία που έχουμε πάντως στην, Πορτογαλία, στην Πορτογαλία δεν συμβαίνει τόσο πολύ, αλλά σε πολλές άλλες χώρες ναι, το δεύτερο σώμα έχει συμβουλευτικό ρόλο, άρνηση κυρίας, πάυσης κάποιων διαδικασιών. Αυτό είναι το προφίλ των παρεμβάσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Είτε σαν σύμβουλοι που λένε προσοχή, όπως είναι ο ρόλος της Βουλής των Λόρδων στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι και αυτή αρμοδιότητα των κοινοβουλίων όταν υπάρχει ένα σύστημα με δύο σώματα ή τρία. Εγώ δεν το βλέπω αυτό να έρχεται σε αντίθεση με το συνταγματικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Και έρχομαι τώρα στην επικουρικότητα. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον ορισμό του καθηγητού Μπερνίτσε που εκφράστηκε πάρα πολύ καλά και από την Μεσέντες Μπρέσο ότι δηλαδή η επικουρικότητα είναι μία αρχή που δεν έχει μόνο μία κατεύθυνση, υπάρχει μια αμοιβαιότητα εδώ. Γι' αυτό και πριν από 17 χρόνια όταν έγραψα κάτι για το φεντεραλισμό και για την αρχή της επικουρικότητας, χρησιμοποίησα μια διατύπωση ουδέτερη, αλλά πολύ ουσιαστική πιστεύω. Optimal territorial. Δηλαδή ότι η επικουρικότητα είναι για να μας οδηγήσει στην καλύτερη εκδοχή. Δεν είναι ότι είναι το εθνικό, το περιφερειακό, το τοπικό επίπεδο. Όχι, λέει ότι πρέπει να γίνεται στο επίπεδο εκείνο όπου είναι πιο αποτελεσματική η επικουρικότητα. Δεν λέει ότι όλα πρέπει να γίνονται στο χαμηλότερο δυνατόν επίπεδο ή όλα στα ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Όχι, Λέει ότι κάθε φορά πρέπει να βρίσκουμε το πιο σωστό επίπεδο, το πιο αποτελεσματικό επίπεδο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό για να απαντήσω και στην Ταϊάννα James που συνεισφέρει επικοδομητικά με την παρέμβασή τη, όταν λέει ότι η επικουρικότητα ουσιαστικά είναι ε, σαν να βρίσκεται κανείς ε, κάτω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποταγή, δεν είναι αλήθεια αυτό. Γιατί δημιουργήθηκε η ενιαία αγορά. Και οι ίδιες χώρες που έχουν ε, αυτούς τους νόμους θα πρέπει να τους αντικαταστήσουν με κάποιους άλλους και όταν θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τη θέλουν την εσωτερική αγορά. Οπότε αν συνεχίσουν να τη θέλουν θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν τους ίδιους κανόνες. Σίγουρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δραστηριοποιηθεί πολύ. Θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση, γιατί αν δεν υπάρξει εναρμόνιση δεν θα υπάρξει ενία αγορά. Άρα δεν είναι θέμα υποταγής, είναι θέμα επικουρικότητας. Αν έχετε ευρωπαϊκού μεγέθους αγορά, πρέπει να έχετε κοινού αγώνες, γιατί τότε δεν είναι μία αγορά. Όπως είδατε, τις ερωτήσεις τις διατυπώνω ανοιχτά ακριβώς γιατί βασιζόμαστε στις απαντήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Από τη συζήτηση εδώ για μένα είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να είμαστε πολύ ανοιχτοί στην πράσινη κάρτα. Είδαμε ότι όλοι την υποστηρίζουν και ευχαριστώ και για τις ιδέες σας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για συγκεκριμένα θέματα και όχι γενικά. Η Επιτροπή θα το μπορούσε να βοηθήσει σε τέτοιες συζητήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια εβδομαδιαία συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο επίσης είναι κάτι, ένα συγκεκριμένο θέμα για τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Οπότε πολύ χαίρομαι για τη σημερινή συνάντηση. Και πάλι ευχαριστώ τις εθνικές αντιπροσωπείες που ήρθαν για τις προσπάθειές τους και για τη συνεισφορά τους που ήταν πραγματικά ουσιαστική και βοηθάει πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε εδώ έγκαιρα και πιο νωρί θα έλεγα, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Θα συνεχίσουμε την έκθεση του Παόλο Ράντζελ ο οποίος προφανώς και θα λάβει υπόψη του τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.